και περνάμε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. Θα ακουστεί δήλωση της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζων Κλωτιούνκερ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε με τον συνήθι τόνο για το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν των γεγονότων που πολύ σωστά καταδικάσατε κι εσείς, που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί στο Πακιστάν. Δεν είναι όμως καθόλου δύσκολο εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλήσω για την απονομή του βραβείου του Καρλομάγνου. Είμαι ο ίδιος ε, δύο φορές έχω τιμηθεί μάλιστα το 1980 από τον λαό του Λουξεμβούρου, εκ μέρους του λαού του Λουξεμβούρου έχω τιμηθεί ε, με το βραβείο του Καρολομάγνου και το 2006 προσωπικός. Η σειρά λοιπόν των τιμηθέντων με το βραβείο Καρλομάγνου, με το πρόσωπό σας κύριε Πρόεδρε, συνεχίζεται με τρόπο ιδιαίτερα τιμητικό. Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασία της Νέα Επιτροπής, θα ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι είχα την εντύπωση κατά την προεκλογική εκστρατεία όπου ήσασταν φιλικός αντίπαλος, για να το θέσω έτσι, ότι θα έπρεπε να δώσουμε μια νέα εκκίνηση στην Ευρώπη. Αυτή την εντύπωση είχα αφού επισκέφτηκα 20 περίπου χώρες και 33 ευρωπαϊκές πόλεις. Γι' αυτό ξαναγάπησα την ε, Ευρώπη γιατί καταλαβαίνετε ότι σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα είναι δύσκολο να επισκεφτεί κανείς τόσους τόπους και να συναντήσει τόσους διαφορετικούς ανθρώπους. Είχαμε συμφωνήσει κατά τη διάρκεια σύστασης της νέας Επιτροπής ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε επί της ουσίας, δηλαδή τα βασικά ζητήματα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που σκιαγράφησα στις 15 Ιουλίου και στα τέλη Οκτωβρίου. Όλοι συμφωνήσαμε ότι όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη δεν αποτελούν ε, προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της επικουρικότητας και να επιληθούν τα προβλήματα ανάλογα με το επίπεδο εξουσίας. Δηλαδή, οι τοπικές αρχές μπορούν να δώσουν μία λύση στα προβλήματα που τίθενται σε αυτό το επίπεδο στην Ευρώπη. Με βάση αυτές τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάσαμε τέσσερις από τις 52 πρωτοβουλίες et qui οι οποίες έπρεπε να συζητηθούν. Αυτό το κάναμε λαμβάνοντας υπόψη τις ε, μεγάλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγάλη προτεραιότητα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρό μας, αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Γι' αυτό Τρεις εβδομάδες μετά την ε, θέσπισή της, η Επιτροπή πρόθεσε ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο εξάμεινο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδέθηκε με εμάς την εξέταση αυτού του κειμένου. Λάβαμε υπόψη αυτές τις νέες λοιπόν πρωτοβουλίες που ανέρχονται στις 452. Ε, Όπως ξέρετε, για το 2015 θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα εργασίας για το 2015 αποκλειστικά. Και όχι αυτό που θα αφορά την πενταετή θητεία μας. Περιορίσαμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ασυνέχειας που υπήρχε, γι' αυτό θα αποσύρουμε και θα τροποποιήσουμε και θα αλλάξουμε 83 κείμενα που βρίσκονται επιτάπητος, για τα οποία θα πρέπει να νομοθετήσουμε. Πέρα από το επενδυτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα επενδύσεων, υπάρχουν και τα προγράμματα φορολόγησης και δημοσιονομικών θεμάτων. Όπως σας είπα, τους έξι πρώτους μήνες θα προβούμε σε μία οδηγία σε σχέση με τις ανταλλαγές απόψεων, τις ανταλλαγές πληροφοριών εκεί όπου χρειάζεται. Η Επιτροπή λοιπόν θα υποβάλει ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης, λαμβάνοντας υπόψη ότι εκεί όπου αποκτώνται κέρδη, εκεί θα πρέπει και να φορολογούνται. Και θα ήθελα να πω εντελώς φιλικά ότι μέρα με τη μέρα με καλούν να κάνω αυτό που είπα. Αυτό ακριβώς θα γίνει για το 2015. Όπως είχα πει, θα ήθελα να συγχαρώ τον Φρανς Τίμερμανς για τον τρόπο που συντόνισε τις εργασίες της Επιτροπής για το πρόγραμμα εργασίας, συνάντησε όλους τους επιτρόπους και προετοίμασε αυτό το πρόγραμμα εργασίας με το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να πω ότι είναι αξιέπαινη η προσπάθειά του και γι' αυτό ακριβώς θα δώσω το λόγο στον πρώτο Αντιπρόεδρο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα εργασίας και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο τώρα έχει ο Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμαντς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ εσάς, όπως έκανε και ο πρόεδρος, το βραβείο Καρλομάγνου είναι ιδιαίτερα προσφυλές και σε εσά και σε μένα, γιατί εμείς είμαστε από την περιοχή του Καρλομάγνου. Η κεντρική περιοχή είναι η πόλη του Άχεν, η οποία συνδέεται πάρα πολύ με τις προσπάθειες που έγιναν να επουλωθούν κάποια τραύματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βέβαια το να τιμηθεί κανείς με αυτό το βραβείο είναι ένα από τις υψηλότερες τιμές που μπορεί να λάβει κάποιος Ευρωπαίος. Τα συγχαρητήρια λοιπόν και από εμένα. Θα ήθελα μέσω ημών κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο για την ε, συνεισφορά του στην προετοιμασία του προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015. Όπως είπε και ο πρόεδρος μας, θέλουμε να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες και να είναι όλες για το 2015, όχι για τα έτη που έπονται. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και κάποιες προτεραιότητες για τα επόμενα έτη μετά το 2015, όμως αυτά θα τα διαβάσετε στα προγράμματα εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε η δική μας Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας παραδώσει κάποια κάποιο νέο τρόπο συνεργασίας, το οποίο μπορούμε να κάνουμε μόνο όμως αν συνεργαστούμε στενά με εσά και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν απευθύνει και μια πρόσκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας το χρησιμοποιήσουμε ως μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των δικών μας θεσμών και ας έρθει και ο τρίτος νομοθέτης στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται και αυτό ως Συμβούλιο να παίξει το ρόλο του. Έχουμε 23 νέα μέτρα στον κατάλογό μας. Και πρέπει να σας πω ότι δεν θα ακολουθήσουμε την τακτική του να παριθμούμε κάθε μία δράση μήπως και μας κατηγορήσουν ότι δεν είμαστε πλήρεις. Θα μιλήσουμε μόνο για τα όσα σκοπεύουμε να κάνουμε το 15 τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Ε, όχι πως δεν θα ξεκινήσουμε προετοιμάζοντας και κάποιες ναι. μελλοντικέ ε, εργασίες για τις κατευθυντήριες γραμμές για το 16 και 17, για παράδειγμα πολιετές ε, δημοσιονομικό πρόγραμμα, ενδιάμεση αναθεώρηση κτλ. Και βεβαίως θα σας τηρούμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις. Η πρώτη μας προτεραιότητα όμως, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι να παραδώσουμε το όσο υποσχεθήκαμε στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και θα κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση του προγραμματός μας ε, που θα ακολουθήσει τα όσα έγιναν τον πρώτο μήνα ε, μετά που αναλάβαμε. Έχουμε λοιπόν και τα χρήματα, τα κονδύλια ε, για τα επόμενα τρία έτη και πρέπει να σας πω πως εκεί πολλά θα κάνουμε όπως επίσης και στην ψηφιακή αγορά. Θέλουμε μια σφριγιλή ψηφιακή αγορά. Πώς θα το κάνουμε. Έχουμε το περιβάλλον ρύθμισης για τις τηλεπικοινωνίες, θέλουμε πιο εξυγχρονισμένους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πιο εύκολες πωλήσει και αγορές ψηφιακά, ε, θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε κάποιες διατάξεις στην προστασία του καταναλωτή και πρέπει να σας πω πως μετά από αυτό το θέμα που ακολουθεί είναι η ενεργειακή ασφάλεια, ο ενεργειακός αναφοδιασμός στην Ευρώπη. Και μέσω αυτών θα προωθήσουμε βεβαίως και την πράσινη τεχνολογία. Θέλουμε την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Αυτό είναι σημαντικό για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και μαζί με τα σχέδιά μας να έχουμε ε, ε, μία ένωση κεφαλαίων θέλουμε να προσελκύσουμε τους επενδυτές στην Ευρώπη. Να ενθαρρύνουμε παράλληλα όμως και τον κοινωνικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε δικαιοσύνη και ευκαιρίες για όλους στην κοινωνία μας και θα ψάξουμε να βρούμε νέους τρόπους να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε όλοι οι πολίτες και κυρίως οι μακροπρόσωμα άνεργοι και οι νέοι να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, να έχουν τα προσόντα που χρειάζονται και να μείνουν σε αυτή την αγορά. Θα παρουσιάζουμε ένα πακέτο μέτρων για να προωθήσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων και θα στηρίξουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση των διαφορών επιδομάτων που ε, παρέχονται. Φορολογική δικαιοσύνη. Το ζητούν οι πολίτες. Θα πρέπει τα κέρδη των επιχειρήσεων να φορολογούνται εκεί που έχουν αποκτηθεί. Ακόμα και στην ψηφιακή οικονομία. Θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο δράσης σχετικό μαζί με προτάσεις για την διαφάνεια των φορολογικών αποφάσεων και θα επακινήσουμε τις ε, ε, τις διάφορες προσπάθειες που γίνονται για, τον κοινό εταιρικό φορολογικό συντελεστή. Μετανάστευση. Τι περιμένουν από εμά οι πολίτες. Καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης ε, προς την Ευρώπη, αλλά να είμαστε ένας ελκυστικός ε, τόπος για όσους έχουν ταλέντο και προσόντα και θα δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε ε, στην, ε, για τη στήριξη των δημοκρατικών αλλαγών στους κανόνες που έχουμε. για παράδειγμα, περισσότερη διαφάνεια στις συναντήσεις μας με τα εμπλεκόμενα μέρη και θα χαρώ να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο στο συγκεκριμένο σημείο αυτό. Τα σχέδιά μας τα εξετάσαμε από πολύ κοντά. Θέλουμε να δούμε τι θα προσφέρουμε. Αν δίνουμε προσθέμενη αξία, ας πούμε, στις θέσεις εργασίας και στην απασχόληση σε αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη. Πώς βοηθάμε εμείς χωρίς να δημιουργούμε επιπλέον εμπόδια και φραγμούς. Αναρωτηθήκαμε για όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, αν όντως εμπίπτουν με τις 10 προτεραιότητες, τις οποίες συμφώνησε με το Κοινοβούλιο όταν ε, εξελέγει ο πρόεδρος Γιούγκερ. Επίσης αναρωτηθήκαμε το ίδιο για το κατά πόσο είναι απαραίτητο, χρήσιμο από τις 400 τόσες προτάσεις που εκκρεμούν, που βρίσκονται μπροστά σας, να τις προωθήσουμε όλες. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικής ασυνέχειας που υπάρχει και βρίσκεται και στο συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των δύο θεσμών. Πολύ συχνά παρουσιάζεται ως κάτι που πρέπει να εξασφαλίσουμε, αλλά σε πρακτικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο αυτή η αρχή ε, να εφαρμοστεί και το ε, ανακάλυψα και εγώ τις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα που θα ξεκινήσει ο νέος νομοθετικός κύκλος θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο έτσι ώστε το χρόνο και την ενέργειά μας να τον επενδύσουμε στις προτάσεις οι οποίες πραγματικά θα έχουν επιπτώσεις στην απασχόληση και που όντως έχουν πιθανότητες να εγκριθούν στο άμεσο μέλλον. Οπότε θα εξετάσουμε όλες τις προτάσεις εγκάρσια για να δούμε ποιες θα κρατήσουμε, ποιες θα τροποποιήσουμε και ποιες θα αποσύρουμε. Θέλουμε αποτελέσματα ε, γρήγορα και όπου δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ε, με τρόπο που θα εξυπηρετεί τους στόχους μας θα προσπαθήσουμε να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Για παράδειγμα, η οδηγία για την ενεργειακή φορολόγηση. Εμείς προτείνουμε να την αποσύρουμε γιατί την έχει ε, χαλαρώσει τόσο πολύ ε, το Συμβούλιο που ουσιαστικά δεν έχει πλέον νόημα με τον τρόπο που πέρασε από το Συμβούλιο δεν περιορίζει ε, τις ε, ε, εκπομπές ε, άνθρακα. Επίσης, θέλουμε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση ε, στα οικονομικά θέματα. Θέλουμε και αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ. Μετά μπορείτε να μου φωνάξετε ότι αυτά που δηλώνω είναι ντροπή, αλλά αν με ακούσετε μπορεί να μην χρειαστεί να πείτε κάτι τέτοιο. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως η κυκλική οικονομία αντιμετωπίζεται ως κύκλος ολόκληρος και όχι ως ημικύκλιο. Δηλαδή, μιλάμε για τα απόβλητα και την πρόταση που έχουμε να αποσύρουμε εκεί γιατί θέλουμε να κατεβάσουμε μια νέα πρόταση το 2015 η οποία θα είναι καλύτερη γιατί θέλουμε εμείς να είμαστε στην εχμή ε, του δόρατος έτσι ώστε όταν οι προτάσεις και εμφανιστούν έτσι όταν έχουμε την δυνατότητα να κατεβάσουμε επενδυτικέ προτάσει, αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Αν λοιπόν αποσύρουμε το πακέτο για τα απόβλητα, το κάνουμε γιατί θέλουμε κάτι πιο φιλόδοξο στο τραπέζι. Και θέλουμε εμεί να συνεισφέρουμε με τρόπο που θα προωθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία εκεί που τη χρειάζεται. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε εάν ευθυγραμμιστούμε με το σχέδιο Γιουγκέρ, το πιστεύω βαθύτατα. Εντάξει, δεν θα μου φωνάξετε πω θα έπρεπε να ντρέπομαι. Πολύ ωραία. Αυτέ οι πιο φιλόδεξε προτάσει θα παρουσιαστούν για να προωθήσουμε την οικονομία και θα, θα τα παρουσιάσουμε του χρόνου. Παράλληλα, θα προωθήσουμε τι επενδύσει στου κλάδου μέσω του νέου ε, μηχανισμού, όπω επίση και των διαστρωτικών και επενδυτικών ταμείων τη Ευρώπη πολιτικές και διευθυντήριες γραμμές. Είπαμε πως θα εξετάσουμε και το πακέτο ε, για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Είναι καλές οι προοπτικές, αλλά η μεσοπρόθεσμη πρόταση θα πρέπει ε, να εγκριθεί ε, σύντομα για να κλείσει το κενό που υπάρχει, που είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία μας. Η πρόταση για τις οροφές, για τις εθνικές εκπομπές ήταν τελικά ε, εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και είναι πολύ διαφορετικά αυτά που θεωρούν αποδεκτό αποτέλεσμα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν μέσα στις τρέχουσες ε, διαπραγματεύσεις θα παρουσιάσουμε μια τροποποιημένη πρόταση που ελπίζουμε θα γεφυρώσει το χάσμα αυτό, που θα απηχεί καλύτερα τις συνέργειες που έχουμε με τα πακέτα για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια και θα μειώσει και το διοικητικό βάρος. Και είμαστε αισιόδοξοι. Πώς θα πετύχουμε στις διαπραγματεύσεις, πώς θα συμφωνήσουμε. Και το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για οποιοδήποτε συμβιβασμό σε σύγκριση με τους στόχους που είχαμε θέσει. Όχι, αλλά εμείς ε, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθήσαμε να συμβιβαστούν τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη έτσι ώστε σύντομα να έχουμε καθαρότερο ατμοσφαιρικό αέρα στην Ευρώπη. Έχουμε μιλήσει πολύ για την οδηγία για την άδεια μητρότητος. Να είμαι ξεκάθαρος. Ε, τα φράγματα αυτή τη στιγμή στην πρόσφαση των γυναικών ε, στην αγορά εργασία και στι προαγωγέ αυτών ε, μα απογοητεύουν όπω σα απογοητεύουν και εσά. Λόγω των προτάσεων που έχουμε κάνει πολλές χώρες έχουν καλύτερες, προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες για την άδεια μητρότητα. Αλλά θέλουμε περισσότερε γυναίκε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στην αγορά εργασία. Θα συνεργαστούμε μαζί σα και με το Συμβούλιο να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να απεμπλοκάρουμε την οδηγία αυτή. Εάν όμω. δεν καταφέρουμε μέσα σε έξι μήνες και είμαστε ακόμα σε αδιάξοδα, θα την αποσύρουμε και θα παρουσιάσουμε μια νέα πρωτοβουλία που θα αντιμετωπίζει τους στόχους μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε, ναι, θα παραμείνουμε φιλόδοξοι. Ναι, θέλουμε η οδηγία αυτή να πετύχει. Αν όμω εξακολουθεί να είναι στο δρόμο για το πουθενά θα αναλάβουμε νέε πρωτοβουλίε για να σπάσουμε αυτή τη γυάλινη οροφή που θα επιτρέψει στι γυναίκε να ανέβουν πιο ψηλά στην αγορά εργασία. και θα είναι πιο χρήσιμο για όλου. να επενδύσουμε χρόνο και προσπάθεια σε αυτή τη συζήτηση και να μην συνεχίσουμε με αυτό το ατέρμονο θεσμικό αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή πιέζονται και τα τρία θεσμικά όργανα του επόμενου έξι μήνε να δώσουν μια δυναμική που θα προωθήσει αυτή την πρόταση. Αν το νοείτε θα προχωρήσουμε. Εάν δεν γίνεται θα κατεβάσουμε μια καινούρια πρόταση. Και αυτό στα πλαίσια του νέου κανόνα για την καλύτερη νομοθεσία. Επίσης, καλύτερη και πιο εύκολη εφαρμογή της νομοθεσίας. Εμείς πιστεύουμε πως κάποιες πρωτοβουλίες για την καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει εμείς να κάνουμε μια πιο σωστή αξιολόγηση κυλιόμενη των ε, νομοθετημάτων που παρουσιάζουμε έτσι ώστε οι νόμοι αυτοί να καλύπτουν τους στόχους τους αλλά με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Τι θα ακολουθήσει λοιπόν. Εμείς θα συζητήσουμε τις προτάσεις προς απόσυρση μαζί σας. Και αυτό θα, ε, και η απόσυρση θα αποφασιστεί μόνο αν ακούσουμε και αφού ακούσουμε την άποψή σας. Γιατί ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε είναι οι τρεις εταίροι οι συνομοθέτες να συμφωνήσουν για τις πρωτοβουλίες ε, ε, τις δικές μας. Με χαρά θα συνεργαστούμε και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Θέλουμε να δουλέψουμε μαζί, να εντοπίσουμε τους φακέλους όπου θα μπορούσαμε εμείς να αναλάβουμε την συστράτηση, να προχωρήσουμε γρήγορα, έτσι ώστε σύντομα, το συντομότερο δυνατό να βρέψουν τα αποτελέσματα τα ευνοϊκά οι πολίτες. Δηλαδή, βαθύς, δομικός ε, διάλογος μαζί σας την Άνοιξη και το καλοκαίρι. Αν τα καταφέρουμε, ίσως καταλάβουμε καλύτερα τον τρόπο που πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας στο μέλλον. Και τα τρία όργανα. Βεβαίως το πρόγραμμα το δικό μας, δεν είναι το τέλος μιας διαδικασίας, είναι απλά η αφετηρία. Μέσω διαλόγου και θα χαρώ πολύ να επιστρέψω στις αρχές της επόμενης χρονιάς, αν μου το επιστρέπετε και εσείς κύριε Πρόεδρε, να γυρίσω, να τα ξαναπούμε, να ξανασυζητήσουμε. Σήμερα κάνουμε μια αρχή. Θέλουμε τη στήριξή σας και η Ευρώπη χρειάζεται εμάς, γιατί θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα για πολίτες που θέλουν ανάκαμψη, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τίμερμαν. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ο κύριο Σάιερ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ μαζί με του συναδέλφου να σα συγχαρώ για το σημαντικό βραβείο Καρλομάγνου. Είμαστε στην ε, περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, διακοσμούμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και έχουμε κάνει πολλές φορές συζήτηση για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα σε περίοδο χριστουγεννιάτικη. Και πάντοτε χρησιμοποιούσαμε την έκφραση ότι πρόκειται για μια σειρά προτάσεων που μοιάζουν με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που γεμίζεται με στολίδια. Όμως τώρα βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Βλέπουμε προτάσεις συμπυκνωμένες και ουσιαστικές και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, έχουμε καλές προτάσεις και καλά αποτελέσματα αρκεί ο καθένας να προσπαθήσει να βάλει και τη δική του μπαλίτσα και να γεμίσει με στολίδια το δέντρο. Τουλάχιστον όχι από το ΕΛΚ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στις βασικές προτεραιότητες και αρχές του προγράμματος Juncker για, το, για την προσεχή περίοδο τα ίδια πιστεύω βλέπει και το Κοινοβούλιο ως πρόθεση. Όλοι θέλουμε την ε, διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου ο καθένας με το δικό του το λιδάκι. Πολλές φορές ζητούμε να μπουν και άλλα ζητήματα μέσα, ε, χάνοντας όμως τη λέξη προτεραιότητα, η οποία προτεραιότητα, priority στα αγγλικά, έχει μέσα της, ενέχει μέσα της τον όρο πρώτος. Γι' αυτό λοιπόν προτεραιότητα μπορεί να είναι μόνο μία. Δέκα προτεραιότητες έστω 23 προτεραιότητες και 452 πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικό εγχείρημα και ε, επιλογές. Εμείς για αυτές όλες θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στα κύρια ζητήματα και να αποφύγουμε πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είναι άκρως απαραίτητες. Θέλουμε επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση. Πολύ συχνά το Κοινοβούλιο, οι συνάδελφοι ζητούν να ε, συμπληρωθούν οι προτάσεις με άλλα στοιχεία και νομοθεσία ακριβώς γιατί δεν υλοποιούνται όσα έχουν προγραμματιστεί. Γι' αυτό λοιπόν θέλω ιδιαίτερη εστίαση στα θέματα της υλοποίησης. Θέλουμε ένα πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχευση την ανάπτυξη, περισσότερε θέσει εργασία, κινητικότητα στην αγορά εργασία, καλύτερη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση παντού και όχι μόνο στο χώρο τη πληροφορική, ε, μια εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί απρόσκοπτα με ασφάλεια και, προμήθεια, και οικονομική προμήθεια της ενέργειας, ασφαλής και ενωμένη ψηφιακή αγορά, λιγότερη γραφειοκρατία σε κάθε στάδιο, ε, είτε αυτό είναι το εθνικό είτε αυτό είναι το στάδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, καταπολέμηση της φοροαρπαλλαγής και της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ένα περιβάλλον ε, ε, θετικό, γιατί δεν χρειάζεται ο μικροεπιχειρηματία αρνητικό περιβάλλον, χρειάζεται ευχερή πρόσβαση στο κεφάλαιο και του επενδυτές Και βεβαίω είμαστε υπέρ, κυρίες και κύριοι, τη αλλαγή. Αλλά αυτή η αλλαγή θα πρέπει να ε, κριθεί με βάση την υλοποίηση του Προγράμματος τη Είμαστε υπέρ ενός New Deal, όπου η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από κοινού μπορούν να προσδιορίζουν τις προτεραιότητες. Ελπίζουμε ότι αυτό το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Ελπίζω να δικαιωθούμε στο μέλλον όταν θα χρειαστεί να το κρίνουμε εκ των αποτελεσμάτων του. Προς το παρόν σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ για τη μεγάλη αυτή τη τιμή του βραβείου του Καρλο που λάβατε και που τιμά εσάς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά με αυτό το γνωμικό Προωθήσαμε και την εκλογική μας εκστρατεία το Μάιο, όμως το κοινοβούλιο αυτό διαφέρει από τα προηγούμενα. Είναι το πρώτο το οποίο εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής υπό ένα νέο πνεύμα. Αυτά δεν τα λέω εγώ, το, τα είπατε εσείς κύριε Γιούνκερ κατά την ομιλία σας του Ιουλίου και συμμερίζομαι αυτά που είπατε. Ο τρόπος εκλογής αλλάζει την οπτική γωνία και του Κοινοβουλίου. Δηλαδή ζητούμε μια άλλη σχέση εμπιστοσύνης που διαφέρει από την προηγούμενη. Περισσότερο διάλογο, περισσότερη, ε, περισσότερη διάλογο, περισσότερη ανταλλαγή απόψεων και φυσικά και απόδοση λογαριασμών. Καλύτερη συνεργασία και ε, συχνή επαφή των συννομοθετών. Μια νέα μέθοδο εργασίας μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου μέσω επικοδομητικού διαλόγου. Κύριε Τίμαρμανς, αυτά είχατε πει. Δεν τα λέω εγώ και συμμερίζομαι τα όσα προείπατε. Λυπάμαι γιατί θα πρέπει να σε πω εξ ονόματος της ομάδας την ε, απογοήτευσή μας και το θυμό μας θα ήθελα να σας ε, διαβιβάσω, διότι σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, το πρόγραμμα αυτό δεν ε, συνάδει με τα λόγια που προείπατε. Μοιάζει με λόγους του παρελθόντος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι, ελλείψεις και μία απόδοση στόχων. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν υφίσταται πλέον μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και δέχομαι αυτά που είπατε σήμερα, διότι δεν πρέπει μόνο να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, αλλά και κατά διαφορετικό τρόπο. Θα το προσπαθήσουμε κατά την επόμενη πρότασή μας. Η ομάδα μου έχει προτεραιότητες, τις γνωρίζετε πολύ καλά, μείωση της ανεργίας ιδιαίτερα και ιδιαίτερα για τους νέους. Και όπως σας είπα, θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς το καθεστώς φορολόγησης. Είπα αυτή την άποψη η Επιτροπή υπέβαλε μια σαφή πρόταση. Θέλουμε περισσότερα και θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουμε στον τομέα της φορολόγησης το 2015. Επίσης, το κοινωνικό, τα κοινωνικά πρότυπα θα πρέπει να μας απασχολήσουν για να μειώσουμε τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτή την έννοια Χρειάζεται θετική επικουρικότητα αλλά και μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση που να ξέρει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Γιατί η ομάδα μου έχει ορισμένες επιφυλάξεις. Θα πρέπει να κρατήσουμε τους στόχους μας αν και θα πρέπει να αλλάξουμε τη μεθοδολογία ως προς την άδεια ε, μητρότητας και την συστημική και συστημικούς κινδύνους της οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκερέρο, ο κύριος Συγκλέσιας ε, παρακάλεσε να δοθεί ευκαιρία να σας ε, υποβάλει μια ερώτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκερέρο. Θα ήθελα με τώρα που σας άκουσα να σας ρωτήσω αν νομίζετε πως ήταν σωστό να υπερψηφίσετε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τις προτάσεις τους. Θέλω να σας πω πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο ειδών συμμαχίες. Η θετική συμμαχία, η οποία και ο θετικό συνασπισμό προσπαθεί να δώσει μια απόκριση στις προσδοκίε των πολιτών και να βοηθήσει τα προβλήματά τους και η αρνητική, ο αρνητικό συνασπισμό που θέλει τη σύγκρουση χωρί να προτείνει λύσει. Εγώ θέλω να συνεχίσω με αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν στο να λύσουμε τα προβλήματα. Εσείς θέλετε να είστε με τους εξτρεμιστές που δεν έχουν λύση να προσφέρουν στους πολίτες. E Εκ μέρους της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Φόρτ. Η κυρία Φόρτ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα ξεκινώντας ε, την ομιλία μου να κάνω μια δήλωση για τα συγκλονιστικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Πακιστάν. Εμεί οι γονεί θέλουμε τα παιδιά μα στο σχολείο για να μάθουν και είμαστε βέβαιοι ότι είναι ασφαλή εκεί. Ή θέλουμε να είμαστε, είμαστε στο πλευρό των γονέων αυτών που έχασαν τα παιδιά τους σήμερα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις, η οικονομία μας υφίσταται πιέσεις, οι πόροι παιδια του υφίσταται μεγάλε προκλήσει, η ασφαλεία μα υφισταται πιέσει, οι ποροι μα υφισταται πιέσει, η ασφαλεια μα υφισταται πιέσει και η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Κύριοι και κυρίες Επίτροποι, μιλήσατε για αλλαγή. Πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα σε αυτές τις υποσχέσεις. Χρειάζεται να κάνουμε οικονομικές επιλογές. Βεβαίως και έχουμε υψηλές προδιαγραφές ε, στην ε, οικονομική ευημερία, το περιβάλλον, ε, την ασφάλεια. Χρειάζεται όμως η οικονομία να έχει την προτεραιότητα. Κάθε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περνάει από την εξή απλή δοκιμή. Θα διευκολύνει ή θα δυσχεράνει την ευημερία για τις επιχειρήσεις. Έχουμε δει στο παρελθόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγει νέα νομοθεσία χωρίς να κοιτάει τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή στις νέες επιχειρήσεις, στις μικρές επιχειρήσεις, την καινοτομία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και οι αποφάσεις θα πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Είχατε υποσχεθεί κύριε, κύριε Γιούγκερ ότι θα αναζητήστε και επιστημονικό σύμβουλο από την ομάδα μας. Παρακαλώ αυτή την υπόσχεση να την τηρήσετε. Ε, αν υπάρχουν λοιπόν κάποια δεδομένα ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα ένα νέο νομοθέτημα, έστω αλλά αν δεν υπάρχουν, αν είναι ακριβώς αντίθετα τα δεδομένα και τα στοιχεία, τότε πρέπει να αλλάζει. Μιλήσατε για την ε, κατάργηση της γραφειοκρατίας, θα το κάνετε αυτό. Μιλήσατε για την ε, ανάπτυξη, την αγορά ενέργειας, τις υπηρεσίες, αυτά όλα με μείωση του κόστους, ώστε να βοηθήσουν την ανάπτυξη. Αυτές είναι οι αλλαγές που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Το 2015 θέλουμε να έχουμε το βλέμμα στραμμένο προς το 2050 και όχι προς τη δεκαετία του 50 του 1950. Θέλουμε ψηφιακές αγορές με στοιχεία και δεδομένα που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και που θα ενισχύουν και το εξωτερικό εμπόριο. Εάν δεν επιτέχει η ε, συμφωνία η Διατλαντική Συμφωνία με τις ΗΠΑ για το εμπόριο θα έχουμε μείνει πίσω. Θα χάσουμε επενδύσεις, επενδύσεις οι οποίες στηρίζονται στο ιδιωτικό ε, χρήμα και όχι μόνο στο δημόσιο. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στο δημόσιο χρήμα για τις επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κοινωνικές πολιτικές βεβαίως και πολιτικές για την απασχόληση, αλλά όχι κεντρικές, γιατί το να ξεπεράσουμε τις αρμοδιότητες και να υπερκεράσουμε τις αποφάσεις των εθνικών κρατών και κυβερνήσεων ε, θα φέρει περισσότερα ακόμα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να περικόθουν ε, οι δαπάνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Πρέπει να περικοπούν οι δαπάνες και καθώς είναι τόσο εκτεταμένο το δίκτυο των δημοσίων δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών δομών ε, βρίσκεται ο λαός μας ε, στην υποχρέωση να μεταναστεύει. Πρέπει να επικοινωνήσουμε και με τα άλλα κράτη για να αναζητήσουμε τα ζητή, τους, ε, τις αιτίες της μετανάστευσης και να βρούμε λύσεις για το πρόβλημα της μετανάστευσης τόσο προς όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει αυτό να το δούμε μαζί με τις επιχειρήσεις και να διευκολύνουμε την, τις συναλλαγές όχι με μια γραφειοκρατική και μονολυθική προς, προσέγγιση η οποία θα οδηγεί σε στασιμότητα την οικονομία, όχι με τη γραφειοκρατία, όχι με τις υπερβολικές ρυθμίσεις. Αυτές είναι οι θέσεις μας και θα συνεργαστούμε με όσους τις συμμερίζονται. Ευχαριστώ, κύριε Φόρντ. Ο κύριος Λάιχτφριτ έχει μπλε κάρτα για σας. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι εδώ. Μπροστά. Σας άκουσα μεγάλη προσοχή κυρία Φόρτ. Ένα σημείο με ενδιαφέρει πολύ από την ομιλία σας. Είπατε ότι πρέπει να έχει την προτεραιότητα η οικονομία, οι όμιλοι δεν πρέπει να περιορίζονται στη δράση τους. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεν θα υπάρχουν κοινωνικά δικαιώματα, δεν θα υπάρχουν ε, δικαιώματα των εργαζομένων, θα είναι όλο και χαμηλότεροι οι μισθοί, θα συμπιέζονται όλα τα, ε, όλα τα ωφέλη για τον εργαζόμενο. Απαντήστε παρακαλώ σε αυτό. Και επίση θα ήθελα να πω, σε απάντηση τόσο είπατε ότι από την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να υποφελούνται οι πάντε και όχι ορισμένοι και ολίγοι. Παρακαλώ. Το να μοιραστούμε τα θετικά και τα πλεονεκτήματα τη ανάκαμψη είναι πολύ σημαντικό και τη ανάπτυξη, αλλά πρέπει πρώτα να πετύχουμε την ανάπτυξη και μετά θα δώσουμε καλύτερε συνθήκε διαβίωση. Και γι' αυτό στηρίζουμε και εμεί κάποιε εκκλήσει για μια πιο στοχευμένη προσέγγιση που θα σέβεται παράλληλα και την επικουρικότητα. Das Wort hat jetzt für die liberale Fraktion. η κυρία Yes, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας εγχαρώ εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για καλύτερη νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου αυτό θα σήμαινε και διαφάνεια. Ε, και περισσότερη εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Αλλά νομίζω η συζήτηση σήμερα γίνεται με βάση ένα έγγραφο το οποίο διέρευσε στον τύπο. Αυτό μου φαίνεται μια μάλλον ασυνήθις διαδικασία. Εγώ θα ήθελα ε, να απλουστευτεί η διαδικασία, να είναι πιο εύκολη, αλλά εμείς πιστεύουμε πως πρέπει να γίνεται μια ευφυής προσπάθεια και όχι με το τσεκούρι να πάμε να ρίξουμε όλο το δέντρο. Δεν θα πρέπει να τα πετάξουμε όλα μαζί, να κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά γιατί θέλουμε καλύτερη νομοθεσία και να αποσύρουμε ό,τι πρόταση υπάρχει μπροστά μας. Βεβαίως και θα πρέπει ε, να περικόψουμε την ε, άχρηστη ε, νομοθεσία, αλλά πώς κρίνουμε τι είναι άχρηστο ή δεν είναι απαραίτητο. Εμείς θεωρούμε στους φιλελευθέρους πως η ισότιμη μεταχείριση είναι πολύ σημαντικό ε, θέμα. Αλλά για εσά η οδηγία κατά των διακρίσεων είναι άχρηστη γραφειοκρατία. Εμείς θεωρούμε στου φιλελεύθερου πω είναι πολύ σημαντική διαφάνεια. Αλλά εσεί λέτε πω ο νόμος για την πρόσβαση στα έγγραφα θα πρέπει να καταργηθεί. Οι φιλελεύθεροι θέλουν και πιστεύουν πω η βιωσιμότητα είναι μεγάλη προτεραιότητα. Αλλά εσεί που θα περικόψετε τη γραφειοκρατία θέλετε ε, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για τα απόβλητα να αποσύρετε τα πακέτα. Εμεί θεωρούμε πω οι δημοκρατικοί κανόνε και το κράτος δικαίου είναι πολύ σημαντικό θέμα και σε πολλά κράτη-μέλη δυστυχώς είναι και θέμα επικαιρότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω δεν προτείνει κανένα μέσο. Και η δημοκρατία ε, και το κράτος δικαίου σας φαίνονται πως είναι περιτά. Επίσης, ε, για ε, το θέμα με τα δεδομένα. Εσείς το αφήνετε πίσω ε, χωρίς ε, να παρουσιάζετε κάποια δικαιολογία. Εμείς πιστεύουμε πως θα πρέπει οι διαδικασίες να ενισχυθούν και όχι εσείς απλώς να γνωρίζετε τα αποτελέσματα του δημοκρατικού διαλόγου. Εμείς πιστεύουμε πως θα πρέπει να αποσυρθούν φάκελοι μόνο και μόνο επειδή τα κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και παραλύει το Συμβούλιο. Μόνο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποσύρονται. Και ξέρετε πως αν απλώς ε, δεν πιέζαμε τα θέματα, δεν θα είχαμε ούτε για τις τράπεζες, ούτε για τα ε, διπλώματα βρασιτεχνίας, ούτε για το άσυλο, ούτε για την εσωτερική αγορά κανόνες. Βεβαίως τον αποσύρουμε κάποιους κανόνες χρειάζεται να γίνει. Αλλά για παράδειγμα, τι θα γίνει με τα φορολογικά κίνητρα που δίνουν τα κράτη-μέλη, τι θα γίνει με την ε, ε, υπερβολική γραφειοκρατία, πώ θα εξασφαλίσετε εσεί πω τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν καλύτερα το κοινοτικό δίκαιο. Και κυρίω θα έχουμε ρήτρα κατάργηση ε, σε όλε τι νομοθετικέ σα προτάσει. Και τέλο, θα αυξήσετε τα επίπεδα πρόσβαση στα έγγραφα και τη διαφάνεια, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη λογοδοσία που κατά τη γνώμη μας είναι και το κλειδί για να έχουμε καλύτερη νομοθεσία. Ξέρετε πως όταν διοριστήκατε κύριε Τίντερμαντς είπατε πως η Ευρωπαϊκή αυτή Επιτροπή γεννήθηκε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν επειδή το είπατε θέλουμε κι εσείς να συνεργάζεστε χέρι-χέρι μαζί μας, να μειώσουμε το ρυθμιστικό βάρος αλλά παράλληλα να εξασφανίζουμε δημοκρατική και διάφανη ε, διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους τη Ενωτικής Αριστεράς η κυρία Κάρη. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή θέλει να ακολουθήσει μία νέα οδό. Δηλαδή, δεν θέλει να μας παρουσιάσει περισσότερο από το ίδιο, από αυτό που είχε προϋπάρξει, αλλά θέλει να έρθει σε καλύτερη επαφή με τους πολίτες. Αυτό δηλαδή που έχει σημασία είναι να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις αλλά να μην αφαιτήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό είναι το πρώτο στο μέλημά μας, δηλαδή να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων έτσι ώστε να μην τα αφαιτούν οι επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε εκ του μηδενός οι πολίτες θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο, να αποτελέσουν το κεντρικό μέλημά μας. Ευχαριστώ εκ μέρους της ομάδας των Πρασινών, ο κύριος Λάμπερτς. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Η νομοθεσία αυτή είναι η νομοθεσία της τελευταίας ευκαιρίας εδώ στην Ευρώπη. Αν θέλουμε λοιπόν να συμφιλιώσουμε τους πολίτες με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα πρέπει να προσεγγίσουμε την Ευρώπη στον πολίτη. Αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει η Ευρώπη μας να εργαστεί για την πλειοψηφία των πολιτών και όχι για μία μειοψηφία. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τρεις άξονες. Καταρχήν κοινωνική δικαιοσύνη. Χρειάζεται να έχουμε ένα τριπλό αλφα στον κοινωνικό τομέα. Μπορεί πολλοί να πούν όμως ότι ο κοινωνικός τομέας δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα αυτό ισχύει πρωτίστως. Μιλήσατε για την φορολογική δικαιοσύνη. Και τουλάχιστον βρισκόμαστε στην καλή, στη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως μέχρι την πλήρη φορολογική διαφάνεια έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Πιστεύουμε επίσης, και δεν το άκουσα αυτό να το λέτε ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Τίμερμανς, αντίθετα με αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί θα πρέπει να ξαναδούμε το οικονομικό πακέτο, να μειωθούν οι ανισότητες, να μειωθεί η φτώχεια, να λάβουμε υπόψη τον περιβαλλοντικό παράγοντα, γιατί οι επιλογές των κυβερνήσεων θα πρέπει να οδηγήσουν στη μείωση των ανισοτήτων και όχι στην αύξησή τους. Επίσης δεν άκουσα να μιλάτε για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Θα πρέπει αυτό το εξάμεινο να αντιμετωπίσουμε το θέμα τους, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου. Ως προς την περιβαλλοντική αηφορία, αηφορία ακούω εδώ και στο Συμβουλίο ότι η μετάβαση αυτή αποτελεί ένα άχθος, μεγάλο άχθος. Όμως θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να προωθούμε την ενεργειακή αυτάρκεια, διότι προς το παρόν εξαρτόμαστε από την αλλοδαπή. Επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσει ο δημοκρατικός άξονας. Υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Άκουσα για διαφάνεια, αλλά το ευρωπαϊκό εξάμεινο που θα πρέπει να έχει κύριο μέλημα τη σύγκληση δεν προωθεί αυτό το στόχο. Θα πρέπει να δώσουμε νομιμότητα στις συζητήσεις και στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων δεν θα πρέπει να λυθούν όλα στα παρασκήνια μεταξύ ανωτέρων υπαλλήλων, διότι ούτε οι μεν ούτε οι δε δεν έχουν να λογοδοτήσουν δημοκρατικά. Δηλαδή τα μέτρα δεν θα πρέπει να επιβάλλονται χωρίς να λογοδοτεί κανείς ε, πολιτικά. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Κύριε, κύριε Λάμπερτς, έχω μια παράκληση. Πάτε πολύ γρήγορα για τους διερμηνείς. Μα ξέρετε, είναι ο ενθουσιασμός της νιώτης, κύριε Πρόεδρε, με καταλαβαίνετε. Τέλος, το θέμα της ε, καλύτερης ε, ρύθμισης. Better regulation σημαίνει no regulation πολλές φορές. Μας είπατε πολλά και ενδιαφέροντα για το θέμα των αποβλήτων. Θα ήθελα να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν πρόκειται για απόσυρση των μέτρων για την ποιότητα του αέρα διότι στο θέμα του REFIT δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το REFIT είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το σώμα αυτό για να αποδυναμώσει τα μέσα κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας. Κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί οι πλέον ευάλωτοι θα πρέπει να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το REFIT δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε απορρίθμιση Επίσης, με εξέπληξε το ότι χρειάστηκαν πέντε μέρες ε, για, την, για τον Επίτροπο Χιλ για να αντιδράσει τη, στην επιστολή των ε, τραπεζιτών για να αποσύρει την οδηγία για τα hedge funds. Θα έπρεπε να έχει αντιδράσει άμεσα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ενθουσιώδης πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, γιατί αυτή η οδηγία έτσι κι αλλιώς έπρεπε να αποσύρθει. Αυτό ήταν σίγουρο. Κύριε Λάμπερτς, ο κύριος Βούλφ θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Mr. Lambert, you suggested... Προτείνατε κύριε Λάμπρεχτ στην αρχή της ε, παρουσίασης πως ο κύριος Τίμερμαντς αντιμετωπίζει αυτή την τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη να στηρίξει τους πολλούς και όχι τους λίγους. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή φροντίζει μόνο τους ολίγους. Εκούτε... Ακούστε με. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος και είμαι μηχανικός. Οπότε κυρίως κοιτάω νούμερα. Κοιτάω λοιπόν λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη και το τι έχει συμβεί από την αρχή της κρίσης. Ποιοι οικονομικά τα πάνε καλύτερα και ποιοι τα πάνε χειρότερα. Αν δείτε λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, γενικά ένα με 2% του πληθυσμού είναι σε καλύτερη θέση ή καλύτερα και οι υπόλοιποι ζουν είτε όπως ζούσαν είτε χειρότερα, είτε με αβεβαιότητα. Άρα λοιπόν οι πολιτικές που ε, ακολουθήσαμε στην Ευρώπη μετά από τις επιταγές της εθνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στο να στηριχθούν κάποιες μειοψηφίες. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των Ελευθεριών και των Δημοκρατικών, ο κύριος Φαράζου. Κύριε Γιούγκερ, ήρθατε εδώ με την επιτροπή σας να μας παρουσιάσετε ένα νέο πρόγραμμα εργασίας, αλλά βλέπω ότι πολύ σας ε, απασχόλησαν οι δημόσιες σχέσεις. Προσπαθήσατε να ξαναδιαμορφώσετε μια νέα εικόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ένα νέο σύνθημα, νέα αφετηρία για την Ευρώπη. Μια χαρά τα καταφέρετε, μα κάθε πέντε χρόνια αυτό το έργο βλέπουμε, να μας δώσετε πίσω τα λεφτά μας. Είδα και στον Περλεμό μπροστά ένα μεγάλο μια πολύ μεγάλη γιγαντοαφίσα με, ε, με το πρόσωπό σας και τον λοιπόν, Team Juncker, ομάδα Juncker. Έχει πέντε πρώην πρωθυπουργού αυτή η νέα επιτροπή. Τέσσερι πρώην ε, υπουργού, δέκα εννέα πρώην υπουργού, επτά πρώην επιτρόπου και μπορεί να έχει και κανέναν δυο νέου ε, ίσω, αλλά φαίνεται σαν να βλέπουμε να επανέρχονται οι παλιοί για να μας ξαναπέξουν το ίδιο έργο της εσωτερικής πολιτικής. Στην ίδια αυτή η επιτροπή, στις οποίες είχεστε εσείς κύριε Γιουνκέρ. Μη φανταστεί κανεί ότι αμφισβητώ τι ικανότητέ σα. Ασφαλώ και όχι. Είσαστε πάρα πολύ καλό. Είσαστε πολύ ικανό στο να κάνετε τη δουλειά σα σωστά. 400 τόσε ήταν οι πολυεθνικέ οι οποίε μπόρεσαν να ξεφύγουν από πολλά δισεκατομμύρια φόρου ε, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, βάζοντα την έδρα του στη φορολογική στο Λουξεμβούργο, στην περίοδο που ήσασταν εσεί πρωθυπουργό και του δώσατε τι ευλογίε σα. Και αυτέ οι επιχειρήσει ασφαλώ θα μα πούνε ότι είσαστε πολύ ικανότερο ε, από των προκάτοχών σας. Αλλά σας παρακαλώ μη μας λέτε σας και και νέοι. 19 χρόνια πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. Επικεφαλής της Ευρωζώνης, Ευρωομάδας. Είστε μια επιτροπή η οποία είναι το ίδιο μοχλιασμένη και το ίδιο, ε, ε το ίδιο κατακάθι έχει όσο ένα παλιό κρασί, μπουκάλι με κρασί. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Επίτροπε, δεν καταλαβαίνω πού το πάτε και τι θέλετε να πείτε. Ωραία ακούγονται τα λόγια σας βεβαίω. Μας είπατε σήμερα, κύριε Τίμερμαν, ότι θα έχετε μια μινιμαλιστική προσέγγιση για την νομοθεσία. Όπως και ο κύριος Γιουνκέρ. Ασφαλώς είστε πολύ πιο ευφυείς, πολύ πιο έξυπνο, πιο μάγκας από όσου προκατόχου ε, έχουν προηγηθεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα μας λέτε να ρίξουμε λίγο λαδάκι στο πιάτο για να, να βουτάμε το ψωμί μας μέσα στο εστιατόριο. Αυτό θα είναι η ρύθμιση που θα επιβάλλεται, όπως η ιστορία με το μέγεθος ε, του τουρσιού αγκούρι ή όποιου άλλου αγκουριού μας είχατε τα προηγούμενα χρόνια. Και πρέπει επίσης να πω ότι όταν, όταν προσπαθήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιολογήσουμε τον όγκο των νομοθετημάτων που επεβάρναν τις επιχειρήσεις μας, μετρήσαμε το 2005 2.000 και σελίδες. 20.000 και σελίδες. Ίσως τώρα να έχουν φτάσει και στις 250.000. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, κύριε Τίμερμαντς, μινιμαλισμό δεν θέλουμε. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο με το τσεκούρι πρέπει να αρχίσετε να κόβετε δεξιά και αριστερά τα περιτά νομοθετήματα, ιδιαίτερα αυτά που επιβαρύνουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί η οικονομία δεν μπορεί να διατηρήσει τα ίδια επίπεδα για τον κάθε έναν, όπως βέβαια για τις αγαπητές ε, πολυεθνικές. Ο μινιμαλισμός σε κάποια σημεία βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο ένας, είναι, το ένα, ο τομέας είναι η διαπραγμάτευση για το θέμα της μετανάστευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είπατε κύριε Γιουνκέρ ότι η ελευθερία των λαών είναι μια διαπραγματεύση, μια αξία. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και βέβαια το άλλο το αδιαπραγμάτευτο είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε λοιπόν μήπως τελικά και τα δύο πρέπει να φύγουν. Και γι' αυτό θα έλεγα πολύ προσεκτικά να κοιτάξουμε τα επόμενα πέντε χρόνια εάν η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ και αν η Βρετανία θα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως αυτά τα πέντε χρόνια να σας απασχολήσουν ακριβώς αυτά τα δύο θέματα. Κύριε Βουλευτά, η κυρία Μπρεσό έχει ερώτηση για σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τον ε, κύριο Φάρατζ κατά πόσο ξέχασε πέρα από τις ρυθμίσεις του Λουξεμβούργου να ρωτήσει κατά πόσο και η χώρα του έχει καρποθεί από αυτές τις ρυθμίσεις. Βλέπω επίσης ότι δεν έχετε πια τη Βρετανική σημαία και αυτό με ευχαριστεί. Και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζετε ίσως ότι εδώ βρίσκεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος γιατί με ρωτήσατε και ποιο ήταν το θέμα, αλλά τουλάχιστον έτσι έχω χρόνο να μιλήσω κι άλλο. Τώρα, για τους κανόνες του Λουξεμβούργου, εγώ το ξεκαθάρισα. Δεν επικρίνω ιδιαίτερα εδώ τον κύριο Γιούγκερ γιατί πιστεύω στη φορολογική, στο φορολογικό ανταγωνισμό και να κάνει κάθε κράτο αυτό που πιστεύει με διαφορετικό τρόπο το οποίο είναι υγιέ για την Ευρώπη. Και μια διόρθωση. Έχετε δίκιο. Δεν έχω σημαίακι πάνω πάνω ε, στο τραπεζάκι μου, αλλά δεν είχα ποτέ αγγλική σημαία, είχα πάντα τη βρετανική, το Union Jack. Νομίζω ότι η μάχη της Παντιέρας έπεσε θύμα των μαχών του πολέμου του Βελγίου. Για να δούμε λοιπόν το επόμενο. Στην επόμενη Ολομέλεια θα έχετε τη Union Jack. Union Jack έτσι. Εσείς είσαστε για τις, ε, μάχη της Παντιέρας. Uh, Κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη σύνοδο στραφήκατε κατά μια ομάδας η οποία επεδείκνυε σημαίες ή σημεία τα οποία κατηγορούσαν για ρατσισμό κτλ. Και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα επικρίνατε τις εθνικές σημαίες που είχαμε πάνω στα έδρανά μας. Εγώ έψαξα τον κανονικό τον κανονισμό εντωμεταξύ. Στο 15ο παράρτημα του κανονισμού εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται ότι απεικονίσει συμβόλων είναι ανεκτές εφόσον δεν είναι προσβλητικές ή δυσφημιστικές. Η λέξη λοιπόν ρατσιστής και ομοφοβικός είναι όντως δυσφημιστικές. Αν και θα περίμενα ε, κάτι περισσότερο από την ε, αριστερή ομάδα, δεν θεωρώ ότι είναι όλοι τους εκεί ρατσιστές και ομοφ... οι δυσφημιστές καλύτερα. Εσείς θέλετε να πείτε ότι η Union Flag, η Βρετανική σημαία είναι είτε ρατσιστική είτε δυσφημιστική, υβριστική. Όχι, δεν είναι υβριστική. Απλώς διαπιστώνω πως σήμερα δεν έχετε φέρει σημαίακια. Το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Να προβάλλετε τη σημαία σας. Και το έχουμε παρατηρήσει και εγώ και οι προκάτοχοι. Θέλω να πω το εξή ωστόσο. Ε, διαμαρτυρηθήκατε όταν ε, σήκωσαν πλακάτ κάποιοι εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά στην συνεδρίαση των Βρυξελών που αναφέρατε εσείς, Ιταλικό μερίδιο η αντιπροσωπεία της ομάδας σας είχε επίσης σηκώσει πλακάτ. Περίμενα ότι και για τη δική του στάση θα, διαμαρτύρω, θα διαμαρτυρώσασταν. Κύριε Άνεμανς, όχι, όχι, δεν έχετε άλλο πλέον το λόγο, κύριος Άνεμανς. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όχι, θα τα συζητήσουμε επί του κανονισμού μετά, αλλά τώρα έχει το λόγο ο κύριος Άνεμανς. Ο κύριος Άνεμανς. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παραγωρήσω ως Βέλγος γιατί από την σοσιαλιστική απεργία στο Βέλγιο δεν ήμασταν τα μοναδικά θύματα, αλλά και άλλοι ήταν ε, θύματα. Τέλος πάντων, ως ε, υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και ως κριτικός, ε, επικριτικός ε, εκπρόσωπος της χώρας μου, θα θέλαμε να αναφέρουμε τις ε, προτεραιότητες που θα πρέπει να μειωθούν. Ακόμα και όταν ένας ενεργός ανακυκλωτής απορριμμάτων και ως φλαμανδός πολίτης και πολιτικός το υποστηρίζω αυτό θεωρώ ότι το πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής τέτοιας συνεργασίας εδώ πέρα είναι περιττό και θεωρώ ότι μπορούν όλα αυτά να υποκινηθούν από εμπορικές συμφωνίες σε ό,τι αφορά την ε, ενέργεια, τις συμφωνίες από χώρες που δεν μπορούν να ακολουθήσουν θα οδηγήσει σε σπατάλη χρημάτων και τίποτα άλλο. Και αυτό που περιτρανώνεται είναι είναι οι ευρείες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι λογικό το γεγονός ότι καταρτίζεται νομοθεσία γραφειοκρατική στον τομέα, στον τομέα αυτό και ζητείται κι άλλη νομοθεσία πέρα από τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά έχουν προχωρήσει απαράδεκτα πολύ και γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να μην συνεχίσετε να βγάζεται βγάζετε κρατική νομοθεσία. Επειδή θέλουμε να τα κάνουμε όλα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι ήταν η καλύτερη λύση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ο κύριο Ρίδεμαντ για τη διαδικαστικό. Συνάδελφε, ζητήσατε διαδικαστικό. Έχετε το λόγο. Uh, yes, Mr. President. Uh... Ναι, Πρόεδρε, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, οι συνάδελφοί μου της, του Ιταλικού κινήματος των πέντε αστέρων σήκωσαν ε, κάποια μηνύματα που δεν ήταν προσβλητικά. Θέλω να πω ότι ο εσωτερικός κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου σε όλους αμερόληπτα και όλες οι ομάδες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σεβαστές και αντικείμενο αμεροληπτικής ε, αντιμετώπισης στον πρόεδρο. Αυτό σας ρωτάω πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει προσέγγιση αμερόληπτη. Αν προσβλητικά συνθήματα από εκείνα ε, δεν επιτρέπονται και όταν το θέτουμε λέτε ότι μη προσβλητικά ε, είναι εξίσου με μη προσβλητικά ε, μηνύματα δικά μας και έχετε την ίδια αντιμετώπιση με τους που έχουν προσβλητικά μηνύματα φαίνεται δεν αμερόληπτη αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ για την υποδεξή σας. Το λόγο έχει ο κύριος Τσίπ για το, την ομάδα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τη δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλωσορίζω το γεγονός ότι είπε ότι είναι μόνο η αρχή της συζήτησης και όχι το τέλος αυτής. Αντίθετα με αυτά που υπόθηκαν, εγώ δεν θα διατηνόμουν ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παλιά, σκονισμένη και δεν φέρνει καμία αλλαγή δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει σε μια καλύτερη νομοθεσία. Ναι, η αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου είναι αναγκαία. Ίσως έχουμε κάποια επικάλυψη, ίσως να υπάρχουν κάποια κενά τα οποία εμποδίζουν τις δραστηριότητε μας και θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια. Ίσως να υπάρχει δυναμικό που δεν χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Αυτή η αναθεώρηση συνδεόμενη με την μετακύληση κάποιων προγραμμάτων και νομικών πράξεων από την προηγούμενη θητεία απαιτούν γρήγορες αποφάσεις για το πακέτο για τον καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα για τα απόβλητα Φερρυπίν. Και τρίτον, συμφωνώ με τις προτεραιότητες που περιγράψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερα υποστηρίζω την ιδέα της ενεργειακής ενώσεως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η, ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια η άρση των ενεργειακών νήσων, η απερίμωση ε, του εφοδιασμού, ε, ότι δεν θα έπρεπε να προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν προτεραιότητα και εν ώψη της κρίσης στην Ανατολική Ευρώπη. Μετά η εσωτερική αγορά και ο τρόπος της λειτουργίας. Υπάρχει ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αυτό είναι πολύ σημαντικό και η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Και θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε και ευφυή ανάπτυξη και το επιχειρήν πρέπει να υποστηριχθεί κυρίως ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του πακέτου για τις επενδύσεις. Εξίσου πολύ σημαντικό είναι να φορολογούμε τα κέρδη εκεί που γεννώνται, στην πηγή. Ε, πολύ συχνά, κυρίως ε, στην αρχή της μεταμόρφωσης προς την οικονομία της αγοράς, της μετατροπής αυτής σε χώρες όπως η Πολωνία, σε χώρες που υπάρχουν θέματα για τη μεταφορά των κερδών και μετά η κυκλική οικονομία και πώς συνδέεται αυτή με την ε, βιολογική οικονομία όπως αναφέρθηκε στα στρατηγική του 2020. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγκε έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, Πρώτε Πρόεδρε, Επίτροποι, Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι πρέπει να καθοριστούν νέες κατευθύνσεις για την Ευρώπη και να καθοριστεί και ένα νέο επίπεδο φιλοδοξιών. Αν θέλουμε να εστιαστούμε επί ισχυρών ιδεών για την νέα κατεύθυνση για την Ευρώπη, ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η μηχανή που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, δεν λειτουργεί, η παραγωγή θέσεων απασχόληση και θα πρέπει να ξεκινήσει η παραγωγή θέσεων απασχόληση για να ξεπεράσουμε την αποτελμάτιση και ε, να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις κοινωνικές ε, αποκλήσει μεταξύ κρατών μελών και να ανοίξουμε το δρόμο ε, για νέες δραστηριότητες. Πράσινη μετάβαση, ευφυή και καινοτόμο οικονομία επιθυμούμε. Αλλά για να γίνουν αυτά πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Και περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προωθεί ένα νέο πολιτικό μείγμα πολιτικών όπου έχουμε εξυγίανση οικονομική αλλά ύψιστη προτεραιότητα πρέπει να έχει ανάπτυξη που θα έχουμε μεταρρυθμίσεις αλλά μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν το δυναμικό της ανάπτυξης και δεν θα περικόπτουν απλώς τις δημόσιες δαπάνες όπου πάνω απ' όλα θα έχουμε ύψιστη προτεραιότητα για τις επενδύσεις. Αυτό σημαίνει να έχουμε επενδυτικό σχέδιο που είναι σε θέση να υποστηρίξει στατηγικά έργα που λείπουν από την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να έχουμε περιθώριο για επενδύσεις όσον αφορά το οικονομικό κλίμα που θα δημιουργηθεί και το φορολογικό και ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φόροαποφυγής και να αποκλείσουμε επιβλαβή ανταγωνισμό φορολογικό. Αυτό είναι το επίπεδο φιλοδοξιών που περιμένουμε. Να υπογραμμίσω απλώς ότι είναι ιστορικό καθήκον που είναι στα χέρια σας, δηλαδή ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Uh, uh, σας ευχαριστώ. Υπάρχει μπλε κάρτα. Ο κύριος Γιάλ. Κύριε Ροντρίκης μικροφώνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας είδατε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αναφερθήκατε στις παρατηρήσεις σας στη σημασία δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πιστεύετε, θεωρείτε ότι το ευρώ, αυτό το νόμισμα για όλους, πιστεύετε ότι το ευρώ βοήθησε ή εμπόδισε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Το πρόβλημα δεν θεωρώ ότι είναι με το ευρώ. Το ευρώ μπορεί να καταστεί ισχύση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα είναι ότι η Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση είναι ε, ελληματική. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση, θα πρέπει να υπάρχει σωστός συντονισμός για να υποστηρίξουμε τη ζήτηση σε ό,τι αφορά τις χώρες με έλλειμμα και θα πρέπει να έχουμε σωστές ικανότητες. Υπό τους όρους αυτούς θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλη θέση, πολλές θέσεις απασχόλησης και μεγάλη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντούντα για ένα λεπτό. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σήμερα ακούσαμε επανειλημμένα από το στόμα του κύριου Τίμερ μας και της κυρίας Βουλευτού δηλώσεις σημαντικότατες. Σήμερα μεγάλο μας καθήκον στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Είναι ένα αρνητικό φαινόμενο από το οποίο υποφέρουν πάνω απ' όλα οι νέοι. Πρέπει να δημιουργήσουμε προπτικές για τους νέους. Προπτικές που τους επιτρέπουν να ζουν αξιοπρεπώς στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να πρέπει να ψάξουν εργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή δεν είναι καλή λύση είναι κάτι σημαντικότατο. Τον Ιανουάριο του 2014, εδώ και ένα χρόνο μόλις, δημοσίευσε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βιομηχανική αναγέννηση. Και ο, η κυρία Μπινκόφσκα, σήμερα που είναι επίτροπος, τότε ε, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβιομηχανοποίησης της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν κύριε Πρόεδρε να τεθούν τα εξή ερωτήματα. Μιλάμε για ανανέωση βιομηχανική, την αναεκβιομηχάνηση της ε, ε, Ευρώπης. Τι κάνουμε όμως. Μέχρι τώρα τι κάναμε πάνω σε αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς να εξηγήσουμε, πώς να συνδέσουμε μάλλον την ανάγκη αυτή που υπάρχει για την ανάπτυξη με το προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το κλίμα. Το χρόνο αγόρευση έληξε, διακόπτει ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ, έχετε μπλε κάρτα. Ο κ. Κόμπε. Um, Συμφωνείτε μαζί μου. Παρακολούθησα αυτά που είπε η κυρία Ροντρίγκε οι κυβερνήσει δεν δημιουργούν θέσει εργασία. Οι επιχειρήσει δημιουργούν θέσεις απασχόληση, όχι οι Αυτό μπορεί να είναι κάτι καινοτομικό για αυτό το πανευρωπαϊκό ε, την πανευρωπαϊκή σοσιαλιστική αυτή συνέλευση. Αλλά γι' αυτό ο κόσμο θέλει να έρθει στην, ε, για να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, στην Σκοτία, στην Ιρλανδία και όχι για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή αν βρείτε κάποια ερώτηση να απαντήσετε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Πότε επιτέλους θα έχουμε λύσεις βιομηχανικής όσον αφορά την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Πότε θα υπάρξει ένα πρόγραμμα που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, διότι βλέπω ότι είναι ένα μέσο καταπολεμήσεως της ανεργίας, ανάπτυξης της Ευρώπης, και θα τη βοηθήσει αυτό να βγούμε από την κρίση. Αν είναι να δώσουμε χρήματα κάπου, εκεί πρέπει να τα δώσουμε. Και το θέμα ε, ε που, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταλίτσκα. Κύριος Ταλίτσκα είναι επόμενο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση και θα ήθελα να συνεχίσω στα πλαίσια της σοβαρής αυτής συζήτησης. Μας παρουσιάσατε το πρόγραμμα πριν από κάποιες ημέρες ε, για να προετοιμαστούμε. Αλλά αφετέρου ελπίζω ότι οι πληροφορίες ότι το πρόγραμμα αυτό προήλθε από τις υπηρεσίες είναι κουτσομπολιό γιατί αυτό που περιμένουμε είναι πραγματική πολιτική δουλειά. Για το πρόγραμμα το ίδιο τώρα, επιτρέψτε μου. Θεωρώ ότι είναι καλό το έγγραφο, είναι φυσικά ακόμα γενικόλογο και θα πρέπει να δούμε πού θα πρέπει να διευκρινιστεί, αλλά νομίζω ότι αναφέρεται σε μια σειρά θεμάτων. Αυτό που μου λείπει ωστόσο στο σχέδιο είναι ότι κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να αμελούμε και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν καθημερινά τον πολίτη η οικονομική και κοινωνική ατζέντα σίγουρα απασχολεί τον πολίτη, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ενδεχομένω να τονίζονται λιγότερο. Για το επενδυτικό σχέδιο τώρα. Πολύ λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση έχασε την ευκαιρία να συνδέσει τα ωφέλη του επενδυτικού σχεδίου με τις διευθυντικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στα κρατημέλη. Θα ήθελα να υπάρχει μια αιρεσιμότητα με άλλα λόγια σε ό,τι αφορά την καλύτερη ρύθμιση τώρα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό πρώτο για σήμερα, αλλά με απασχολεί το κατά πόσον θα δούμε σύντονα ένα πραγματικό σύστημα. Αυτό μου λείπει από το σχέδιο. Δεν φαίνεται να υπάρχει σύστημα benchmarks, στόχοι και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Τελευταία παρατηρήση, αν μου επιτρέπετε, καταναλαμβάνω ότι βρισκόμαστε στη φάση απόσυρσης νομοθεσίας. Ελπίζω σωστά να κάνουμε, αλλά θα ήθελα αυτή η διαδικασία να βασίζεται σε μελέτες αντικτύπου. Νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες οι επίσης θα πρέπει εκεί να βασίζονται. Δεν είμαι βέβαιος αν σωστά κατάλαβα και πολλοί θα εκτιμούσαν μια διευκρίνηση από αυτού. Μάλιστα λοιπόν, καλή αρχή και κλείνω πρόεδρε. Είναι η πρώτη, το πρώτο βήμα αυτό. Θέλουμε ένα στενερό σύστημα το οποίο θα μας αποφέρει καλύτερη νομοθεσία. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Επόμενος ο ο κύριος Γιουρίστη Αμπάουντς. Μιλάτε για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης Μα ζητάτε να πιστέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν ήταν θέμα πίστη. Μα είπατε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ακούσαμε προσεκτικά αυτά που είπατε και διαβάσαμε την ανακοίνωση. Προσπαθώ να βρω λόγους για τους οποίους θα μπορούσα να πω στους πολίτες της Ευρώπης ότι ε, είμαι ερωτευμένο με το λαό της Ευρώπης. Αυτό είναι εύκολο να το πω, αλλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και του είναι δύσκολο θα πρέπει να εφαρμόζουμε την αρχή της αλληλογγύης αυστηρά. Φοβούμαι όμως ότι για το περιβάλλον εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα κάνει σωστά. όσο μας προαναγγέλουν προγράμματα όλο και πιο φιλόδοξα. Διότι είναι θέμα πίστης. Δεν γνωρίζουμε αυτές τις προτάσεις που είναι τόσο φιλόδοξες και για την αλλαγή την δημοκρατική που λένε ότι θα προαγάγουν. Λένε ότι στοιχηματίζουν υπέρ της διαφάνειας. Το σημειώνουμε, θα δούμε. Αλλά για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών θα δούμε τι χρειάζεται. Χρειάζεται άλλο πρότυπο, άλλη Ευρώπη. Και πρέπει να είναι μέρος αυτών των αλλαγών. Και δεν βλέπω τίποτα από αυτά στο πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Evans, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω και πολλοί συνάδελφοι, και εγώ συγκλονίστηκα την περασμένη εβδομάδα. άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παρατήσει δύο νέου περιβαλλοντικού νόμου για τον καθαρό αέρα και στόχου τη ανακύκλωση. Ε, αυτό στέλνει ένα αρνητικότατο μήνυμα σε εκείνου που περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί όσον αφορά τι περιβαλλοντικέ δράσει. Ξέρω από τη δική μου εμπειρία στην Ουαλία ότι είναι θέματα κρίσιμα για τη δημόσια υγεία και δημιουργούν χιλιάδε θέσει απασχόληση πράσινε. Θα το θεωρήσουμε ως υπόσχεσή σας ότι θα μας δώσετε πιο φιλόδοξες προτάσεις. Θα περιμένουμε ε, ανυπόμονα τις προτάσεις. Ενθαρρύνθηκα όμως ότι είδα ότι συμπεριλάφθηκε ο όρμος ε, στο Swansea για επενδύσεις ε, δεν θα είναι μόνο ανανεώσιμο η πηγή ε, ενέργειας για μελλοντικές γενιές, αλλά θα δημιουργήσει και θέσεις ενέργειας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί νέα τεχνολογία με πραγματική συμμετοχή της τοπικής κοινότητας τέτοιου είδου βιώσιμε επενδύσει για δημιουργία θέσεων απασχόληση πρέπει να βλέπουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πεντιτσίνη, ο κύριος Πεντιτσίνη. Αξιότιμοι συνάδελφοι και εγώ όπως και ο κ. Ντεμπέρτ έχω, επιστημονική, ε, έχω σπουδάσει επιστημονικά θέματα και κοιτάω τα στοιχεία βασικά. Εμόνιση της ατμόσφαιρας πάνω από 400.000 θανάτους πρώιμου προξενεί κάθε χρόνο. Επιτρομή Juncker τι κάνει, αποσύρει το σχέδιο επενδύσεων το πακέτο για τον καθαρό τον σφαιρικό αέρα. Σύμφωνα τι εκτιμήσει τη ίδια τη Επιτροπή, ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε 580.000 νέε εργασίε με αποτελεσματική αποδοτική χρήση των υφισταμένων αρχών ενεργειών, εξοικονομώντα πηγέ ενεργεία που είναι και δαπανηρέ. Η Επιτροπή Juncker τι κάνει, αποσύρει το σχέδιο των επενδύσεων, το πακέτο για την κυκλική οικονομία χάνουμε περίπου 600 εκατομμύρια τόνους υλικού που βρίσκονται στα απόβλητα. Κάθε χρόνο τα χάνουμε που θα μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Αυτά τα υλικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 600 δις οικονομίες το χρόνο. Μειώνοντας εκπομπές του αερίου θερμοκηπίου κατά 2 με 4% το χρόνο. Αλλά η Επιτροπή Juncker τι κάνει. Αποσύρει από το σχέδιο των επενδύσεων την οδηγία για τα απόβλητα στα συστήματα της υγείας ε, έχουμε, ε, γίνονται διάφορες απάτες και επιβαρύνουν τους πολίτες. Τι κάνει, βγάζει το, το, το, χαρτοφυλάκιο για τη διαφάνεια στον τομέα των ιατρικών. Περνάμε φοβερή κρίση οικονομική και οι πολίτες μας ζητούν ελιμοσύνη και οι επιχειρηματίες αυτοκτονούν και ρίχνει χρόνια και χρόνια εργασιών η Επιτροπή Γιούνκερ και εκατοντάδε υπαλλήλου που ετοίμασαν τι προτάσει και, και σπαταλά θάλασσε χρημάτων για μελέτε, αξιολογήσει, απόδοση κλπ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, εμεί ε, δεν είμαστε εχθροί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούμε ότι είναι εχθροί των πολιτών. Εμεί όμω τσακωνόμαστε με εσά, τα μέλη αυτού του κοινοβουλίου που του ψηφίσατε και εξακολουθείτε να του υποστηρίζετε και που δεν τρέπονται για όλα αυτή την... Ε, που δεν εξοργίζεστε μάλλον με όλα αυτά τα απέσια πράγματα τα οποία βλέπετε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Παπαδάκη, για ένα λεπτό. Το μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Κλιμάκωση τη επίθεση κατά των λαών και εργαλείο για την ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων με μόνιμη, ακόμα πιο αυστηρή πλέον επιτήρηση δίνεται πρίκα στα μονοπόλια ακόμα περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις με βασική προϋπόθεση πάνθηνους εργάτες με ελάχιστες ελαστικές εργασιακές σχέσεις. η ενεργειακή ένωση η ενιαία ψηφιακή αγορά το ελεύθερο εμπόριο με τις ηνωμένες πολιτείες και οι άλλες αναδιαρθρώσεις ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις και φέρνουν νέα δεινά στο λαό οι λεγόμενες αγορές δηλαδή το κεφάλαιο ούτε πείθεται ούτε εξευμενίζεται μόνο ανατρέπεται αυτό και η εξουσία του και χρειάζεται σήμερα άμεση λαϊκή παρέμβαση τώρα για να ανακτηθούν οι απώλειες για ζωή χωρίς αγορές ευρωπαϊκή ένωση και μονοπόλια με το λαό πραγματικό αφεντικό στον τόπο του ευχαριστούμε. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, μιλάμε για ένα πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον επόμενο χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ρεαλιστικό. Ευχαριστώ για την προσέγγιση σας και αυτό που ε, προτείνουμε πρέπει να εκτελείται. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αν κάτι δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα για τον επόμενο χρόνο, αυτό σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Δεν θα θέλαμε αυτό το σημαντικό σημείο να εξαφανιστεί. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Και τώρα Κάτι πιο συγκεκριμένο. Ε, μιλήσαμε για την ανεργία. Είναι σημαντικό ο κόσμος να έχει δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα. Στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπω αρκετά σημεία που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση ή να μειώσουν την ανεργία. Το συζητήσαμε. Χρειαζόμαστε ενέργεια φθηνότερη άνοιγμα στην αμερικανική αγορά, ενεργειακό εφοδιασμό ασφαλή. Πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές ενεργειακές πηγές, να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες. Δεύτερη πτυχή, σας ευχαριστώ που το υπογραμμίσατε αυτό. Η ψηφιακή αγορά θα πρέπει να ξεκινήσει ο τριγωνικό διάλογο το ταχύτερο δυνατόν. Θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο. Τρίτο στοιχείο, ο οδικό χάρτη που αφορά τη βιομηχανική μας πολιτική. Χάρη στην επανεκβιομηχάνηση που ήταν ένα βασικό θέμα για την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φτάσουμε ελπίζω σε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα δώσουμε δουλειά στον κόσμο. Ευχαριστώ κύριο Μπούλμαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε της Επιτροπής. Κύριε Αναπληρωτή, Αντιπρόεδρε της ε, Αναπληρωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπατε θα γίνει πιο πολιτική αυτή η Επιτροπή. <clears throat> Το αντίθετο όμως έφερε ότι θα συμβεί. Αυτό για το οποίο συζητούμε σήμερα είναι αν θα πετύχει αυτό. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το πετύχουμε από κοινού αυτό. Το έγγραφο αυτό δεν μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι απόψεις για το πρόγραμμα εργασίας γιατί δεν το έχουμε στη διάθεσή μας ότι αυτό όμως το έγγραφο το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε δεν τα δείχνει επαρκώς όλα αυτά και σε πολύ, πολλές πτυχές δεν ξέρω σε τι οφείλεται αυτό αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και αυτά τα θέματα με ένα παράδειγμα να προσπαθήσω να επεξηγήσω τι εννοώ αυτό το σώμα η Ευρωβουλή κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία πέρασε και πέτυχε στην ρύθμιση των τραπεζών της έκθεσης Κάρας του συναδέλφου μας ότι όλα τα χρηματοοικονομικά ε, ιδρύματα από το 2015, από του χρόνου δηλαδή, ανά χώρα θα πρέπει να αποδεικνύουν πού ποια κέρδη κάνουν και πού ποια, ποιους φόρους πληρώνουν είναι μια καλή αρχή αυτή. Εκεί κάθεται ο συνάδελφος Κάρασα. Άκουσε προσεκτικά. Αυτά τα περάσαμε και τα πετύχαμε για το ΕΛΚ. Εκεί βρίσκεται και ο συνάδελφος Λάμπερτ, ο οποίος ε, πέτυχε αυτά τα πράγματα για τους πράσινους. Και από πλευράς μας, ε, για τους σοσιαλδημοκράτες, ε, τα καταφέραμε. Είναι τόσο απαράδεκτο αν η ομάδα μου σήμερα από εσά αναμένει δεδομένων των συζητήσεων που έχουμε για πρακτικές αποφυγής φορολόγησης επιτέλους να επεκταθεί αυτή η αρχή σε όλες τις πολυεθνικές ε, επιχειρήσεις. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η πρόταση στο πρόγραμμα εργασίας σας σε, μέσα σε μια νύχτα, σε μια μέρα θα διασφάλιζε ότι θα έπαβαν αυτές οι αθέμητες πρακτικές και ότι επιτέλους θα είχαμε δίκαια φορολόγηση για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη παντού λέτε και υποθέτω ότι είναι μια νέα εξέλιξη αυτή, ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα εργασίας λέει μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Θα κατατεθεί και ελπίζω ότι θα υπάρχει αυτό το στοιχείο σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Είναι ένα καλό παράδειγμα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας αν ο ένας αφουγκράζεται τις απόψεις του άλλου και τις σέβεται. Θέλουμε να είμαστε εταίροι. Δεν υπάρχουν όμως μονόδρομοι. Έχουμε φιλοδοξίες και προσδοκίες από την Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Στη συνέχεια Χένκελ ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμά σας πιο πριν από τους εκπροσώπους του ΕΛΚ θεωρήθηκε χριστουγεννιάτικο δέντρο ως ευχολόγιο με δώρα και δέκα κεράκια έβαλε ο αντιπρόεδρος τις δέκα σας προτεραιότητες σε αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πρέπει να πω έχω ένα πρόβλημα με την πέμπτη προτεραιότητα δηλαδή όσον αφορά την νομισματική ένωση. Σε όλους είναι σαφές ε, η παγκόσμια οικονομία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα αυξάνεται περισσότερο από ό,τι η Ευρώπη η Ευρώπη αυξάνεται ταχύτερα από ότι η Ευρωζώνη ίδια. Έχουμε λοιπόν ειδικό ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ευρωζώνη και δεν μπορώ να το αποφύγω. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το πρόβλημα σε σχέση με το... δεν είναι μόνο σε σχέση με τον νότο της Ευρώπης αλλά επίσης και για τη Γερμανία. Μπορούμε να το δούμε αυτό σε σχέση με τους άνεργους νέους στη Νότια Ευρώπη και με τα πλεονάσματα όσον αφορά τις εξηγωγές ε, στη Γερμανία. Πότε θα ε, προσαρμόσουμε τις ανάγκες ε, του ενιαίου νομίσματος ε, στην Ευρώπη και πότε θα αρχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε, αυτούς τους, σε αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις. Ευχαριστώ. Στην συνέχεια, Ντεσαρνές. Κύριε Πρόεδρε, αποφασίσατε να κάνετε πολιτική. Αυτό είναι καλό μαντάτο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι, η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί εκ νέου επί των ουσιαστικών και ήρθε η ώρα. Το ουσιαστικό ποιο είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε μια οικονομία που είναι κοινωνική. Το επενδυτικό σα σχέδιο ακολουθεί σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα θα πρέπει να προχωρήσουμε, να θέσουμε επιτάπητο σε ένα χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης φορολογικής, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον πραγματικά σταθερό για τις επιχειρήσεις και να προχωρήσουμε προς την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Και μετά, εξίσου σημαντικό, δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα, θα πρέπει η Ευρώπη να βρει τη δυνατότητα να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου, το σχέδιο για το κλίμα, κοινή πολιτική για τη μετανάστευση, πραγματικές εξωτερικές πολιτικές και αμήνης. Βλέπουμε σήμερα ποια είναι η κατάσταση στον κόσμο και πόσο είναι επικίνδυνος ο κόσμος, κυρίως με αυτά που συνέβησαν στο Πακιστάν, τα οποία τα σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι, θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί των δύο βασικών ε, τομέων των μεγάλων προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να προχωρήσουμε συγκεκριμένα επί πέντε χρόνια. Μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, να δείξουμε στου συμπολίτε μα ότι η Ευρώπη του δίνει πραγματικά υπεραξία. Όμω ότι θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρώπη ότι πραγματικά υπάρχει. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Παπαδημούλη. Κύριε Γιούγκερ, είναι στο πρόγραμμα της Κομισιόν οι ομές επεμβάσεις στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις των κρατών μελών. Πριν λίγες ημέρες, μιλώντας για την Ελλάδα, υποδείξατε στους Έλληνες να ψηφίσουν τα δικά σας οικία πρόσωπα και να μην κάνουν λάθος. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι δική σας δουλειά. Θα τολμούσατε να κάνετε παραμονές εκλογών μια τέτοια δήλωση για τη Γερμανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα μπορούσατε να σταθείτε ως πρόεδρος της Κομισιόν ούτε 24 ώρες. Πότε αποφάσισε κάτι τέτοιο η Κομισιόν. Με βάση ποια άρθρα των συνθήκων. Ακούστε, το κόμμα μου ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για λύσεις μέσα στην Ευρωζώνη με ανάπτυξη, με δικαιοσύνη, με βιώσιμο χρέος, με κράτος δικαίου, με ισχυρό κοινωνικό κράτος ακραία δεν είναι αυτή η πολιτική αλλά η πολιτική της τρόικα που εσείς υποστηρίζετε που φέρνει ανεργία ύφεση ανισότητες έκρηξη συνοχής και αποπληθωρισμό. μας υποσχεθήκατε αλλαγές ξεκινώντας αλλά ολοένα και περισσότερο μοιάζετε με δίδυμο αδελφό του κυρίου Μπαρόζο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τίμερμαντς, καμιά φορά είναι καλό να επανεχόμαστε θεμελιώδη και να ξέρουμε γιατί βρισκόμαστε εδώ. Εάν βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε εδώ και πάνω απ' όλα για να όλοι μαζί να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, δηλαδή ενός πολιτισμού που πάντα προσπαθεί να βρει την ισορροπία μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της δυνατότητας για, ε, για τους περισσότερους από εμά να μπορούν να κερδίσουν τη ζωή τους, να ζήσουν άνετα. Λοιπόν, η εξουσία της πρωτοβουλία είναι στα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και σας δίνει μια ευθύνη όλο ιδιαίτερη. Θα δώσετε προνόμιο στο κοινό όφελος των Ευρωπαίων, το ευρωπαϊκό κοινό όφελος, να, στο συμφέρον αυτό να προθείτε. Ποιο είναι αυτό, μονίμως να επιδιώκετε αυτή την ισορροπία μεταξύ του κοινωνικού τομέα, του περιβάλλοντος και της οικονομία. Υπονομεύοντας μέσω υπονομεύοντα το θέμα τη ποιότητα τη ατμόσφαιρα, της κυκλικής οικονομίας και, το, ε, και την εργασία των εγγύων γυναικών υπονομεύεται και αυτή την ισορροπία. Πηγαίνεται κατά τη Ευρωπαϊκή Κοινωνική Σύμβαση Συμφωνία. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα χρόνο να επιστρέψετε, να αναστραφεί αυτή η κατάσταση και να λάβετε ξανά αυτό το κοινό όφελος υπόψη. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή Ο... Η κυρία ο κύριος Λονγκρίν, σα ευχαριστώ πολύ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντα το εξή. Καταρχά να μην ζητώ καρβγάσω. Για τον κύριο Φανρόμπα, ο οποίο παίρνει μια τεράστια σύνταξη, ενώ δεν πληρώνει ουσιαστικά φόρους σε κάτω μέλο. Αυτή τη στιγμή που τα προβλήματα κλιμακώνονται, βλέπουμε ότι ο κύριος Φαρόμπα βγαίνει στη σύνταξη στην πλάτη του φορολογούμενου. Και μιλάτε πλέον για την, την ε, εμπιστοσύνη των πολιτών. Πώς μπορούμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, επιβάλλοντα επιπλέον φόρου, προκειμένου οι πολιτικοί που βγαίνουν στη σύνταξη να έχουν τεράστιε παχυλέ συντάξει και να συνεχίσουν να ζουν με υψηλωτικό βιωτικό επίπεδο εις βάρος των πολιτών. Ένα άλλο σημείο στο πρόγραμμα εργασίας είναι νέα πολιτική για την νέα μετανάστευση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του κυρίου Γιούγκερ. Αυτό θεωρούμε ότι θα έπρεπε να το αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Δεν θα έπρεπε να είναι θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπω πρόκειται να μα επιβάλλεται, να επιβάλλετε στα κράτη-μέλη μια μετανάστευση την οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Δεν έχουμε θέσει εργασία για του κατοίκου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο μάλλον για την ε, νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την μετανάστευση. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει στέγη, δεν υπάρχουν θέσει εργασία για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για πολίτε των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ω συνήθω, ποιο θα πληρώσει τελικά τα σπασμένα, οι εργαζόμενοι. Ποιοι θα πληρώσουν τελικά την τη ροή αποτυχημένων πολιτικών που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω από το 43% των πολιτών δεν πήγαν να ψηφίσουν. Έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη, θεωρώ, οι πολίτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Μποργέζιο έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, στην παρουσίασή σα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ μας παρουσιάσατε περήφανα το σημείο που αφορά την καταπολέμηση της φοραφυγής και την πρόθεση της φορολογικής ισότητας. Είναι παράξενο όμως που σε όλο το πρόγραμμα δεν αναφέρεται τίποτα συγκεκριμένο, ούτε και μια μικρή οδηγία που να δείχνει πώς ε, μπορείτε να καταπολεμήσετε και να προλάβετε ε, αυτές τις ε, ατασταλίες ε, και, και το λαθρεμπόριο ε, το, όπως παραδείγματος χάρη που οδηγούν σε φοροδιαφυγή ε, έναντι ε, των τίμιων πολιτών. Τι κάνετε αγαπητέ πρόεδρε Γιούνκερ. ένα κάτω μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν υπάρχουν τέτοιες, δεν εφαρμόζονται Και είναι στη δική σας χώρα. Στη χώρα σας υπάρχουν προβλήματα. Σας λέω ότι στο Λουξεμβούργο ανοίγεται, θα πρέπει να ανοίξει μια έρευνα. θα πρέπει ο, ε, ο πολίτης παρουσίασε το, το ε, σκάνδαλο αυτό που θα έπρεπε να εμποδιστεί. Ε, και αυτό το σκάνδαλο που ξέσπασε θα έπρεπε να σα εμποδίσει αν γίνεται πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκαλύφθη, συγχαρητήρια. Ο δρόμο πρέπει να ακολουθηθεί πραγματικά πρέπει να είναι διαφορετικό τη απελευθέρωση των χωρών μα από τη φυλακή ε, του ευρώ και να δοθούν στους λαούς μας η νομισματική κυριαρχία και να ελευθερωθούν από τους businessmen ε, και τους εκπροσώπους ε, της ε, Τρόικας, όπως εσείς. Ευχαριστώ. Λεγκρίπ, επόμενος συνάδελφος. Κύριε Λεγκρίπ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Γιούνκερ, τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμανς και θέλατε να επικεντρωθείτε από αυτά που είπατε σε μεγάλους στόχους, κάποιες μεγάλες προτεραιότητες, να επικεντρωθείτε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των ουσιαστικών. Εν ονόμα της γαλλικής αντιπροσωπείας του ΟΕΛΚ θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που φαίνεται για μας τους ευρωβουλευτές, τους Γάλλους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ ότι είναι βασικές προτεραιότητες μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής του ασύλου και της μετανάστευσης και χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή στρατηγική κοινή για την ενέργεια ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Κατά τη διάρκεια του 2015 θα πρέπει να σημειωθούν σημαντικές προόδοι όσον αφορά τους δύο αυτούς άξονες που έχουν προτεραιότητα. Σαν συντονίστρια τώρα του ΕΛΚ και στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών θα ήθελα να επενθυμίσω εντάχει δύο χαρτοφυλάκια σημαντικά. Ε, το πρώτο που είναι προτεραιότητες, μια προτεραιότητες του ΕΛΚ είναι η επόμενη οδηγία γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια θα θέλαμε να καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταθμίζει όσο μπορεί στι διαπραγματεύσει που γίνονται στο Συμβούλιο, ώστε να, το σχέδιο οδηγία για πιο ισχυρή εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια να προωθηθεί. Των μεγάλων επιχειρήσεων των εισηγμένων. Women on boards, όπω λέγεται. Ε, έχουμε καταλήξει στο Κοινοβούλιο ένα συμβιβασμό που είναι ε, πολύ καλό και πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα θα πρέπει τελικά να προωθηθεί και ολοκληρωθεί το 2015 στο σχέδιο οδηγία ε, για τη γονική άδεια Περιμένουμε ε, προόδους ε, ξεκάθαρες, ρεαλιστικές, λογικές, ε, δηλαδή ε, στο εξάμεινο δεν είδαμε να υπάρχει κάποια πρωτοβουλία, δεν ακούσαμε κάτι γι' αυτό. Θα πρέπει να προσέξετε να μην υπάρχει επαναχώρηση σε τον τομέα και να προστατεύετε, ε, να μην γίνει καμία πιστοδρόμηση να αφορά τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας. Μάλιστα σας ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής η κυρία Βίλμοτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και παρουσιάσατε το πρόγραμμα εργασίας κύριε Γιούγκερ στο Κοινοβουλίο. Θα ήταν καλό να το πούμε αν είχε παρουσιαστεί και όχι με καθυστέρηση. Έχοντας ακούσει την παρουσίασή σας έχω κάποιες παρατηρήσεις. Η πρώτη μου παρατηρήση όσον αφορά τους φορολογικούς παραδείσους. Αναγνωρίζω το γεγονός ότι λέτε ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Όμως ε, αυτό θα είχε συμπεριληφθεί διαρωτώνται κάποιοι κοινικοί αν δεν υπήρχαν τα Lux Leaks ως σκάνδαλο. Πέρσι θέλαμε άμεση δράση να αναλυθεί κατά της φοροδιαφυγής τονίζοντας προτεραιότητες όπως ε, εκθέσεις αναχώρα και μαυροπίνακες για εκείνους ε, που φοροδιαφεύγουν. Αυτό είχε γίνει πέρυσι. Μέχρι σήμερα πολύ λίγη δράση είδαμε να αναλαμβάνεται. Σε σχέση με τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζονται οι μειώσεις των μισθών τους, ε, οι υπηρεσίες περικόπτονται μέρα με τη μέρα, κάθε εβδομάδα. Όλοι οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να πληρώνουν τους φόρους τους και βλέπουν το επίπεδο διαβίωσής τους να συστέλλεται και να περικόπτεται και έχουμε ταυτόχρονα άλλους που αποφεύγουν το να πληρώνουν φόρους και να ζουν υπεύθυνα. Χρειαζόμαστε νομοθεσία τώρα, εδώ και τώρα άμεσα. Δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε τα προβλήματα. Δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά το πακέτο των αερομεταφορών. Θα ήθελα να σας για, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Θα υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις για δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ρήπανση 400.000 ανθρώπους σκοτώνει κάθε χρόνο. Τώρα να καταργηθεί νομοθεσία που θα έσωζε τόσες πολλές ζωές δεν είναι μόνο πραγματικά ανησυχητικό, είναι απόλυτα ανεύθυνο. Αποστέτε μήνυμα. Ναι, σας άκουσα κύριε Τίμερμανς εγώ. Ακούστε με κι εσείς. Ε, το να διαγράφετε νομοθετικό έργο που θα ίσως ζητώ σε ζωές είναι ανεύθυνο. Δηλαδή τι μήνυμα στέλνουμε. Ότι δεν ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να προαγάγει προοδευτική πολιτική για το περιβάλλον. Σας ζητώ, απευθύνω έκκληση να επανεξετάσετε αυτή τη θέση σας τώρα, εδώ και τώρα αμέσως κάρτα μπλε υπάρχει για ερώτησή σας. Δεν θα πάρω πολλέ, δεν θα δεχτώ πολλέ τέτοιε μπλε κάρτε γιατί πιέζει ο χρόνο. Διαφορετικά θα έπρεπε να μείνει όλη τη νύχτα εδώ η Επιτροπή μέχρι αύριο το πρωί. Εντάξει, ε, το έχετε συνηθίσει, αλλά εδώ έχουμε και δικαιώματα του ανθρώπου. Κύριο έχετε λοιπόν την μπλε κάρτα. Και μετά η κυρία Βίλμορτ θα απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς ε, την συνάδελφο το εξής σε σχέση με την εκστρατεία που είχε γίνει και τώρα, Ευρωπαίοι που έχουν χαμηλότερο εισόδημα ουσιαστικά ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβουν μια σειρά αποφάσεων που θα παράσχουν νέες προοπτικές για αυτούς τους ε, πολίτες. Δεν θεωρείτε ότι το νέο πρόγραμμα θα έπρεπε να αναζητήσει να διασφαλίζει το ελάχιστο εισόδημα που θα μπορούσε να διασφαλιστεί, ελάχιστο μισθό ως ελάχιστο εισόδημα. Ευχαριστώ μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό συσχετίζεται με αυτά που είπα πιο πριν. Όμως δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να σέβεται όλους τους πολίτες και πρέπει όλοι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και στη συνέχεια η κυρία Τόμασιτς ένα λεπτό. Ο πρόεδρος. Ο Γιούγκερ έχει ένα πάρα πολύ φιλοδοξό πρόγραμμα για την Ευρώπη, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η φιλοδοξία αυτή μα ε, σπρώχνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω να μην ε, είναι παραμύθια όλα αυτά και στο εγγύς ε, μέλλον να μην σκάσει φούσκα αυτή. Θα είναι η πρώτη φορά που δεν, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζει στον χρυσελεφάντινο πύργο της και θα θεωρεί ότι όλα πάνε καλά και όμορφα. Έχουμε πλέον μια καινούργια επιτροπή, ένα καινούργιο πρόεδρο. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν δίκαιο να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Να δράσουν σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Τίμερμανς, ο οποίος μίλησε για το ευρώ, το οποίο θα πρέπει ή την Ευρώπη που θα βελτιώνει και όχι απλά θα παρεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων που θα βελτιώνει τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις όχι απλά θα ε, αυξάνει τη γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά όμως την περισσότερη Ευρώπη που προεξαναγγέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ φοβάμαι ότι θα μας πλήξει αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Βίξτρεμ τώρα έχει το λόγο ευχαριστώ πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρίσκεται εδώ πέρα και που μας παρουσιάζει το έργο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολύ καλό αυτό, αλλά θεωρώ ότι μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη η πρόταση. Καλώς ορίζω ιδιαίτερος το γεγονός ότι η προτεραιότητά σας για την νόμιμη μετανάστευση αναφέρεται και αυτό έχει ω στόχο να καταστήσει την Ευρώπη πιο ελκυστική για ερευνητέ, για φοιτητέ. Αυτά τα χρειαζόμαστε. Για να υπάρξει σωστή οικονομική ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και νόμιμοι και ασφαλείς τρόποι προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να έρχεται εδώ αν ε, απειλείται στην χώρα προέλευσης του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το νεκροταφείο που έχει καταστεί η Μεσόγειος. χιλιάδες άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και χαίρομαι και σε ό,τι αφορά τα, περί, τα θέματα ψηφιακής οικονομίας. Να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιδεικνύει τόλμη και δεν υποκύπτει. σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Φερέρα. Η κυρία Φερέρα, ένα λεπτό. Ο κύριο Φερέρα, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Βλέποντας αυτό το πρόγραμμα βλέπουμε ποιο είναι το νόημα που τόσες φορές έχει αναφερθεί από την Επιτροπή Γιούνκερ. Ένα πρόγραμμα επενδύσεων που θα δίνει λέει δημόσιες εγγυήσεις για ένα τεράστιο πρόγραμμα εταιρικής σχέσης δημόσιας και ιδιωτικής που θα μπορέσει να λειτουργήσει σε μια ε, λογική <clears throat> κερδοφορίας των ιδιωτικών ε, κονδυλίων, των ιδιωτικών κεφαλαίων θα συνεχίσει η ανεργία των νέων. Θα έχουμε περαιτέρω απελευθέρωση των πολιτικών. Είναι συμβολικό το ότι έχουμε χαρτοφυλάκια τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν τις κοινωνικές, ε, τα κοινωνικά θέματα όπως για παράδειγμα τα θέματα μητρότητας και βλέπω μια τεράστια οπισθοδρόμηση σε αυτά τα χαρτοφυλάκια και στο περιβάλλον. Δείχνει εδώ το πρόσωπό της ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι Επιτροπή του Μεγάλου Κεφαλαίου. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χαρτοφυλάκιο των μεγάλων κεφαλαιούχων και των ε, μεγάλων επιχειρήσεων. Άσχετα ποιο κάθεται στην ε, καρέκλα του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκείνοι κάνουν κουμάντο. Όλα είναι παρελθόν και δεν υπάρχει μέλλον. Και αυτό πραγματικά είναι απελπιστικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και στην επόμενη, ο είναι ο κύριος Βόιτ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γιούγκερ μιλήσατε εσείς και κάνατε λόγο σε ένα πρόγραμμα εργασίας ε, με πάμπολες επενδύσεις που θα διασφαλίσουν το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω ένα λεπτό για την ερώτησή μου. Σας ερωτώ καταρχήν πού θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις ώστε να καταπολεμηθούν τα αίτια της μετανάστευσης. Αντί νομιμοποίηση και ολοκλήρωση ασκείται ποιήση στην αγορά εργασίας ε, με 24 εκατομμύρια ανέργους που θα αυξηθούν ακόμη περαιτέρω. Λέτε ασκειται πιεση στην η φοροδιαφυγή θα αυξηθουν ακομα περαιτερω λετε οτι η φοροδιαφυγη θα καταπολεμηθει και η φοροαπάτη. Όμως οι φόροι, είπατε, πρέπει να πληρώνονται εκεί που ε, δημιουργείται το εισόδημα. Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό μετά το πρότυπο που ισχύει στο Λουξεμβούργο. Η φορολογική αυτή η δικαιοσύνη θα ισχύει και για τους εργαζόμενους ή μόνο για τους επιχειρηματίες. Πού παραμένουν οι επενδύσεις στην κοινωνική δικαιοσύνη. Πιστεύετε στις εθνικές διαφορές ε, και ιδιομορφίες στην Ευρώπη με το ενιαίο νόμισμα. Μπορεί το ενιαίο νόμισμα να καταπολεμήσει όλες αυτές τις διαφορές. Ευχαριστώ πρόεδρο. Στη συνέχεια ο κύριος Πρέντα παρακαλώ. Ευχαριστώ απείρως κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι σαν συντονιστή στο ΕΡΚΕΤΑ εξωτερικές υποθέσεις και είμαι πολύ ικανοποιημένο, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακαλύπτω στο πρόγραμμα εργασιών για το 2015 σαν προτεραιότητα την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Είναι μια προτεραιότητα αυτή και για μας. Ήδη το επεξεργαζόμαστε το θέμα. Ο συνάδελφος Edward Κούκαν χειρίζεται το θέμα και Είδαμε πολύ σημαντικό θετικό μήνυμα πλευρά του Επίτροπου Χαν επ' αυτού και είμαι πεπισμένο ότι θα συνεργαστούμε άριστα μαζί, έτσι δεν περαιτέρω, για τα τελευταία χρόνια εξεπλάγημεν κάπω από την αλλαγή στο νότο και στα στην ανατολικά. Μα βρήκε απροετοίμαστου η αλλαγή και καμιά φορά όσον αφορά τι αποφάσει εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε το συνέστημα ότι δεν είμαστε πολύ καλή θέση. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε επίγνωση σήμερα ότι η μεταρρύθμιση της, της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας δεν μπορεί να είναι κάτι απλώς διακοσμητικής φύσεως. Πρέπει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις μεγάλες σημερινές προκλήσεις και θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ Ανατολών και Νότου. Συγγνώμη, Λεπρόεδρο, συνεχίστε. Συγγνώμη που σας διακόψα, Λοιπόν, ήθελα να πω ε, κάποια πράγματα επίσης επί της συμφωνίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες, διότι αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν σημασία ε, ε, για την οικονομική ανάπτυξη, για τις απασχόλησης, αλλά και όσον αφορά την πολιτική. Αυτή η εταιρική σχέση είναι κρισίμου σημασίας για μας και η Ευρώπη θα είναι σημαντικός παγκόσμιος παράγων αν καταφέρει να πετύχει στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς εταίρους. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Μετά η κυρία Τόγια έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ, κύριε Αντιπρόεδρε, Επίτροποι, εμεί εκτιμούμε την αφετηρία, δηλαδή το να σταματήσουμε τι επαφέ με το παρελθόν. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το σημείο θα πρέπει να προχωρήσει ει βάθο, κυρίω όσον αφορά τη σχέση με το Κοινοβούλιο, την πολιτική σχέση. Αν θέλετε πιο ανοιχτή Ευρώπη για του πολίτε, αν προχω... θέλετε να προχωρήσουμε προ την ίδια κατεύθυνση. Από αυτή την άποψη, όπω είπατε, όπως έλεγε ο κύριος Γκερέιρα δεν είμαστε συντονισμένοι. Πρέπει να γίνεται προσπάθεια καθορισμού, ορισμού των διατάξεων και προτεραιοτήτων. Καλύτερη ρυθμίσεις. Θέλουμε better implementation πέρα από το better regulation. Μείωση της γραφειοκρατίας, να μην έχουμε άξιε διαδικασίες. Να χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια να επικρατήσει. Εκείνο που θέλω να πω ουσιαστικά όσον αφορά το περιεχόμενο είναι ότι είναι κεντρική σημασία, αμέσω σημασία η υλοποίηση του σχεδίου των επενδύσεων που έχει και το όνομά σα κύριε Γιούνκερ. Θα ήθελα όμω να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική πολιτική. Δεν θα υπάρξουν επενδύσει και ανάπτυξη αν δεν κάποια πράγματα. Σήμερα το πρωί κάναμε μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά την ευελιξία, την αναθεώρηση των κανόνων και όσον αφορά την υλοποίηση σαν διαφορετική προσέγγιση των κανόνων που ήδη ισχύουν. Θα ήθελα λοιπόν η συζήτηση η πρωινή, αυτά που υπόθηκαν, να αντικατοπτριστούν στι πρώτε πράξει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το έγγραφο για την ευελιξία που περιμένουμε σαν ένα είδο δώρο μετά τα Χριστόγεννα ε, και μιλώ εν ονόματι τη χώρα μου. Το θέλουμε. 40% των εκλογών των Ιταλών εξέλεξαν το κόμμα μου που έκαμε πρόταση. Πιο ισχυρή Ευρώπη, αλλά διαφορετική Ευρώπη. Θέλουμε μια ευελιξία η οποία να είναι ευφυή, δηλαδή χρήσιμη για την επίτευξη του κοινού στόχου της ανάπτυξη. Θέλουμε επενδύσεις, καλές δαπάνες, μια ευελιξία η οποία βοηθά την ανάπτυξη του ΑΕΠ, να μην καταστρέψει τα δημοσιονομικά και να έχουμε μια ευελιξία που οδηγεί σε δαπάνες δημόσιες άχρησης. Θέλουμε ε, ε, επενδύσεις, η χρηματοδότηση προγραμμάτων της Ατζέντα 2020, προγραμμάτων, προγραμμάτων του προγραμμάτους Juncker, των διευθυντικών ταμείων. Η συζήτηση θα πρέπει να επηρεάσει λοιπόν τις πρωτοπράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περισσότερες κοινωνικές πρωτοβουλίες θέλουμε αυτών των τριπλών αξώνων μας άρεσε. Θέλουμε πρωτοβουλίε για τον πολιτισμό, για την κοινωνική οικονομία ε, και για τα διάφορα ιδρύματα και κυρίως συγκεκριμένα ε, σημεία για τον στόχο τον περιβαλλοντικό που ήδη υπενθύμησαν και οι συνάδελφοί μου. Σε ευχαριστούμε. Ο Γκέρικε, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γι' αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 θα έπρεπε να υπάρξει μια νέα αρχή και σας ε, έδωσα, εξέφρασα την εμπιστοσύνη μου γι' αυτό. Αλλά δεν πρόκειται εδώ μόνο για μένα. Τις προηγούμενες εβδομάδες πολύ ήμουνα στην ε, δική μου εκλογική περιφέρεια και είπα στους πολίτες όταν συναντήσω τον πρόεδρο Γιούνκερ τι να του πω, πέντε θέματα θέλω να σας διαβιβάσω πρόεδρε για την ε, εκπαίδευση για τους νέους ε, που κατά τα Χριστούγεννα εργάζονται θελοντικά σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Είπαν να αλλάξετε την πολιτική για τους πρόσφυγες, να βρείτε κοινού κανόνες που θα βοηθούν τους ε, ανθρώπους αυτούς. Ένας νέος με τρία παιδιά μου είπε να με ερημνήσετε για φορολογική δικαιοσύνη, όχι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά για εμάς τους απλούς πολίτες και τις οικογένειές μας. Ένας φούρναρης από τη Δρέσδη είπε ότι η νομοθεσία δεν πρέπει μόνο στις, στα γραφεία σας να εκπονείται. Ας πάνε να μαθητεύσουν οι υπεύθυνοι για το νομοθετικό έργο να μάθουν περί τίνος πρόκειται. Ένας άλλο από το Βερολίνο είπε να δείτε τι γίνεται για τα παιδιά και τις οικογένειες όσον αφορά τον φιλικό προς τις οικογένειες χαρακτήρα της νομοθεσίας. Αυτό θα είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις οικογένειε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια έχετε τον λόγο εσείς ε, Φέντερλαϊ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς Πρόεδρο Γιούγκερ που βρίσκεστε εδώ. Σας εμπιστεύτηκα κατά τις εκλογές ε, της, ε, του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά όταν ακούσαμε ότι το πακέτο για την ποιότητα της, της ατμόσφαιρας και για τα απορρίμματα θα αποσυρθούν, νιώθω ότι προδόθηκε αυτή η εμπιστοσύνη μας. Έχω καινούργιες ελπίδες ε, από εσάς κύριε Τίμερμαντς όταν μας είπατε ότι όλα αυτά θα επενισαχθούν με κάποιο τρόπο, αλλά ξέρετε η υπομονή εξαντλείται και αν δεν υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά τα θέματα, θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερο χάσμα δυσπιστίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, γιατί σας έδωσα την εμπιστοσύνη μας, την εμπιστοσύνη μου και πιστεύω ότι μπορούσατε να αλλάξετε την Ευρώπη για να υπάρξει μεγαλύτερη ευημερία. Αλλά ελπίζω πραγματικά ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην είναι να καταργήσει τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Αλμπιόλ Γκουσμάν. Για ένα λεπτό, η κυρία Αλμπιολ Σας ευχαριστώ κύριε Γιούγκερ. Είπατε ότι είσαστε ερωτευμένος με την Ευρώπη. Σας προσκαλώ να επισκεφθείτε μαζί μου μια κοινωνική μονάδα στη Μελίγια και θα δείτε πόσο αμέσως θα χάσετε αυτό τον, ε, αυτή την ε, ε, σχέση ερωτική και πρέπει να μεταφραστεί το πρόγραμμα σε μια γλώσσα που θα κατανοούν όλοι. Τι είναι πίσω από αυτό το πρόγραμμα εργασίας σας. Το πρόγραμμα εργασία σας αφορά το ελεύθερο εμπόριο με τις ΗΠΑ ώστε οι πολυεθνικές να μπορούν να δρουν όπως κατά το δοκούν όπως επιθυμούν. Περικότερες, περισσότερες περικοπές, φτώχεια, μεγαλύτερη ανεργία. Το φράκινγκ για το σχιστολιθικό αέριο είναι το πρόγραμμά σας για τα κέρδη των πολυεθνικών. Η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών ώστε τα δικαιώματά μας να γίνουν αγαθά και εμπορεύματα. Το σχέδιό σας είναι όλα να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα φορολογικά θέματα του Λουξεμβούργου. Juncker στο Λουξεμβούργο. Νέοι επίτροποι. Ένα δηλαδή πρόγραμμα πρόγραμμα εργασίας ε, για μια πολιτική η οποία θα στραγγαλίζει τον λαό και θα είναι υπέρ εκείνων που ταξιδεύουν στην πρώτη θέση. Το πρόγραμμά σας είναι οι πολιτικές που εμείς θα καταπολεμήσουμε κύριε Γιούγκερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Μπάλτς στη συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά πρόεδρε. Καταρχήν τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Γιούνκερ και τον αντιπρόεδρο Τίμερ μας θέλω να τους ευχαριστήσω που συζητούμε μαζί τους το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το χαιρετίζω ότι αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες χειροπιαστές δράσεις ε, για το πώς θα μπορέσει να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι σημαντικό πιστεύω να τονίσουμε ότι η Ευρώπη πάλι στα κυριότερα θέματα πρέπει να επικεντρωθεί, στα μείζωνα ζητήματα και προβλήματα λιγότερο στα υπουσιοδέστερα. Και θα ήθελα να σας ενδυναμώσω ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ομοθεσία εκβάθρο να την επανεξετάσετε και να έχετε την τέλμη στο τέλος τέλος περί την ομοθεσία να την ε, διαγράψετε, να την αποσύρετε. Αναμένουν οι πολίτες από εμάς πρωτοβουλίες για καλύτερη νομοθεσία. Οι επιχειρήσεις δίκαια και νόμι, θεμητά περιμένουν λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη πρόσβαση, πελασιμότητα σε δυνατότητες χρηματοδότησης Γι' αυτό οι προτεραιότητε αυτές τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα υπόσχονται πολλά ω προοπτική. Δύο προτεραιότητες στον περιορισμένο χρόνο μου θέλω να τονίσω. Πρώτον, νέα προαγωγή για θέσεις απασχόλησης, επενδύσεις, ε, δημιουργία εργασίας. Το πρόγραμμα επενδύσεων εδώ από πλευρά σας είναι ένα σίγουρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη που θα αποκατασταθεί σε σχέση με τους ε, κύκλους των επιχειρήσεων. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σημαντικό εδώ χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις να προαθούν στα κράτη-μέλη, δημοσιονομικές ε, και οικονομικές, ώστε για τη δημοσιονομική διακυβέρνηση να υπάρξει σταθερότητα και ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπέρεση στη συνέχεια που θα λάβει τον λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, το θέμα LuxLeak ε, πέρασε από εκεί και ευτυχώ δεσμεύεστε σήμερα η φορολογία ε, να αποκατασταθεί σε χώρες όπου εκεί που δημιουργούνται ε, τα κέρδη. Αυτό ανακοινώσατε στο πρόγραμμα εργασίας σήμερα. Χρειαζόμαστε περισσότερο φως να ρηχθεί στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσετε όσον αφορά αυτό το δρόμο που για μας είναι απόλυτα ουσιώδης και έχουμε επικροτήσει αυτή την προσέγγιση. Στο ίδιο πνεύμα περιμένουμε επίσης ε, πρωτοβουλίες ούτως ώστε το reporting κατά χώρα να γίνει μια πραγματικότητα, είναι μια διεκδίκηση παλιά του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι σήμερα είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Επ' αυτού δεν ακούσαμε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά το περίφημα better regulation, καλύτερη νομοθεσία, φοβόμαστε, διότι είδαμε ότι αντί να ερμηνευτεί το better regulation και να θεωρηθεί σαν εγκατάλειψη των διαδικασιών των περιπλόκων, ε, θα μπορούσε να γίνει ένα μέσο να αποσυρθούν από την ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κείμενα που, δεν που δυσαρεστούν τη βιομηχανία, προφανώς όπως αφορά τη μόλις του ατμοσφαιρικού αέρα ή της κυκλικής οικονομίας ή κείμενα που θα δυσαρεστούσαν τα κράτη-μέλη και αυτό είναι προφανώς η περίπτωση του κειμένου για την άδεια τη μητρική. Ανακοινώσατε σήμερα ε, νέες ε, προοπτικές και κυρίως μια ανάκαμψη των προσπαθειών για την ε, κυκλική γνωμία, θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι έχετε υπόψη σας για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κάποια δέσμευση συνεργασίας όσον αφορά αυτό το νομοθέτημα που είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε μάλιστα του χρόνου να καταφέρουμε ε, πράγματα στη διάσκεψη των Παρισίων. Ε, αναφέρατε εν παρόδο την αθεώρηση οδηγία των πνευματικών δικαιωμάτων ε, των δικαιωμάτων δημιουργού και θέλουμε αυτό να προωθηθεί ούτως ώστε να μπορεί να ζήσει αυτός ο δημιουργικός τομέας της Ευρώπης και όχι μόνο να ικανοποιηθούν οι ορέξεις κάποιων πολυεθνικών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ιακοβτσίτς, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιούνκε, πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να εκφραστεί εμπιστοσύνη μας σε αυτόν. Είναι μια νέα αρχή αναφέρθηκε. Διαρωτώ με, θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες. Πιστεύω ότι τρεις φάσεις έχουν κύρια σημασία για την εντολή σας. Επενδύσεις, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτή θα είναι η βάση επί της οποίας ή θα επιτύχει ή θα αποτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι για την Οικονομική Νομισματική Ένωση και για την ψηφιακή αγορά που θα ήταν η πέμπτη η ελευθερία, πιστεύω εδώ σε αυτά τα πράγματα. Ακούσαμε πολλές ιδέες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το πρόγραμμα εργασίας θα μπορέσει να δράσει υπέρ των περιφερειών, δήμων και κοινοτήτων και έτσι θα μπορέσει να προαχθεί στο μέλλον και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον. Ε, Ευχαριστούμε. Σπινέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας καλέσω και εγώ να θυμηθείτε αυτά που είπα την Παρασκευή για την ψηφοφορία στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ΣΥΡΙΖΑ καταδίκαζε τους εξτρεμιστές και εκφράσατε τι θέλετε. Θέλετε να δείτε, ε, να βρείτε κάτι διαφορετικό μπροστά σας μου είπανε ότι θα πρέπει να είναι δεξιοσημεία τα πρόσωπα που συνέταξαν τα, το πρόγραμμά σας. Τα πρόσωπα αυτά που οδήγησαν στη φτώχεια την Ευρώπη, στη διάλυση την Ευρώπη. Είναι εκείνοι που αντιλήφθησαν ένα από τα πιο κενά κεφάλαια του προγράμματος. Αυτό για τη μετανάστευση με το οποίο ασχολούμαι εγώ στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Η μετανάστευση τα, θεωρείται με τα γυαλιά τα χθεσινά. Ίσως δεν είδατε ότι έχει αλλάξει το κλίμα, υπάρχει μεταμόρφωση. Σήμερα έχουμε εκείνους πρόσφυγες από τον πόλεμο υπό καταστροφέ κλιματικέ. Έχουμε τη Μεσόγειο που έχει γίνει ένας κοινό τάφος. Χρειάζεται μια αναθεώρηση των κανόνων μας για το άσυλο, ξεκινώντας από το Δουβλίνο 3 που είναι πάρα πολύ αναποτελεσματικό. θα Τελικά κάνει πολλά λάθη τώρα η Ευρώπη και θα πρέπει να μας βοηθήσουν αυτά τα νέα πρόσωπα να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, Φαν Μπρέμπτ, δύο λεπτά. Er ehm, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Αντιπρόεδρο. Από τότε που ανέλαβε τα ενία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Όταν κάνουμε λόγο για την πολιτική για το περιβάλλον, συχνά ακούγεται σαν να είναι μια ενοχλητική πολιτική που ενοχλεί τις επιχειρήσεις, τους πολίτες με γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Θέλω όμως να σας πείσω ότι δεν αληθεύει καθόλου αυτό. Η καλή νομοθεσία που υπάρχουν για την ε, ατμοσφαιρική ρήπανση, για το νερό, για τι υγιεί ε, συνθήκες διαβίωση, ε, μπορούν να φροντίσουν και για πιο πολλέ θέσει απασχόληση, για πιο πολλή κοινοτομία. Αυτό το δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Να σα πω ότι με κάποιου συναδέλφου την προηγούμενη εβδομάδα στη Λίμα είχαμε αυτό το σχετικό έγγραφο και πραγματικά ήταν μια ψυχρολουσία. Προσπαθήσαμε στην Λίμα με δυσκολίε γνωρίζετε άλλωστε και τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο να σημειώσουμε πρόοδο κατά της ε, θέρμανσης του πλανήτη και φαίνεται ότι στις Βρυξέλλες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά έγινε μια ε, μείωση ταχύτητας. Ακούσαμε προσοχή και θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη. Θα ήθελα από πλευρά της ομάδας μας και από πλευρά του Κοινοβουλίου να σας υποστηρίξουμε άκουσα για την κυκλική οικονομία και για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ε, θέλετε να προτείνετε μια νέα πρόταση, να γίνουν τροπολογίες ε, για τις υφιστάμενες προτάσεις, για το θέμα αυτό της κυκλικής οικονομίας και της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Άρα δεν έχουν παραμεριστεί. Θα υπάρξει νέα πρόταση για το 2015 για την κυκλική οικονομία και μια πρόταση τροποποιημένη ή όχι για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το υποστηρίξουμε αυτό, αλλά υπό τον εξή όρο. Να μην μειωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι μας σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία και την ποιότητα του αέρα, της ατμόσφαιρας και το 2015 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορέσουν πραγματικά να στρωθούν στη δουλειά για να είναι πραγματικά βιώσιμη η οικονομία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, επόμενος, επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Χικάτζη Γεωργίου για ένα λεπτό. τη εργασία τη Κομισιόν και πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλη απορία. Απορώ για το μέγεθο ειλικρινά τη κοροϊδία, Η νέα Κομισιόν μα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που φασίζεται στη συνθηματολογία ότι όλα θα αλλάξουν, ότι θα γίνουν νέα πράγματα και νέε πολιτικέ, αλλά στην πραγματικότητα όλα είναι τα ίδια. Διερωτούμε αν διαβάσετε το προηγούμενο πρόγραμμα τη Κομισιόν για να δείτε αυτό που σα λέω βασισμένα σε χιλιοδοκιμασμένες αποτυχημένες πολιτικές πολιτικές που οδήγησαν την ευρώπη και τις χώρες μας στην κρίση και τους λαούς στην εξαθλίωση. τι είναι το νέο όταν οι εξαγγελίες σας για το ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων για τα τριακόσια δεκαπέντε δις βασίζεται απλώς και μόνο στην λεγόμενη μόχλευση δεν είναι και αυτό στην ίδια λογική της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. βαρύγδουπες εξαγγελίες για τα 315 από τα οποία 16 από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 5 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τα υπόλοιπα θα στηριχθούν στου ούτω στους ούτω καλούμενους συντελεστές μόρφευσης. Για να βοηθήσουν ποιου να εξασφαλίσουν σίγουρο περιβάλλον στους επενδυτικούς ομίλους και στα μονοπόλια. Και το κυριότερο θα υπάρξει διαδικασία να πάνε αν θα πάνε αυτά τα χρήματα στις μικρές, μικρές επιχειρήσεις. μια τελευταία φράση κύριε πρόεδρε αν μου επιτρέπετε μου προξενεί μεγάλη απορία οι σοσιαλιστές σας αντιπολιτεύθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο για να σας στηρίζουν κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας. αν αυτό δεν ήταν αστείο... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρος. Επόμενος είναι ο κύριος Φαγιών. Η κυρία Φαγιών, ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε εκατομμύρια Ευρωπαίοι σήμερα δεν έχουν ε, δουλειά. Έχουν χάσει τις αποταμιεύσεις τους. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες ανισότητες και οι προπτικές είναι χειρότερες από ποτέ. Επειδή υπάρχουν και πολλοί από που και πολλές επιχειρήσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή. Η φορολογική παράδειση, η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή, αν συνεχίσουν όλα αυτά μάλλον αν σταματούσαν όλα αυτά θα μπορούσαμε πολλά χρήματα να τα επενδύσουμε στην απασχόληση των νέων, στην εκπαίδευση, στα άδεια της αυροπιλάκια. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία και το ευρύ κοινό θεωρεί ότι είναι κάτι το ανέντιμο η φοροδιαφυγή. Mm. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπόσχονται να καταπολεμήσουν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, αλλά πολλοί υπουργοί στο παρελθόν έχουν παρεμποδίσει όλες αυτές τις ενέργειες. Θέλουμε να υποβάλουν υποχρεωτικές εκθέσεις για τις ε, δράσεις τους, για τις, ε, τους, όλες οι επιχειρήσεις, για να αποτρέψουμε τα φαινόμενα χαμηλής φορολογίας κάποιων εταιριών. Θέλουμε μια δυναμική θαραλέα και ελπίζω σε όλη την Ευρώπη όλος ο κόσμος να δείξει ένα καινούργιο ενθουσιασμό για να διαμορφωθεί η ευρωπαϊκή πολιτική όπως και έγινε πριν από μια δεκαετία. Αν αποτύχουμε, αυτό θα σημαίνει ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από το παρελθόν παρά την όποια φοροδιαφυγή, παρά την άνοδο των ακροδεξιών και της ακροδεξιάς πολιτικής, παρά τους θανάτους στη Μεσόγειο, ακόμα δεν έχουμε βρει συνεκτική πολιτική για την μετανάστευση και το άσυλο. Και ως ε, πολιτικός δεν μπορώ να το υποστηρίζω αυτό. Ευχαριστώ. κυρία Έθριτ, προ την κυρία Φαγιώνα έχει να θέσει μια ερώτηση. Ο κύριος Έθριτ. Αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε με την ανάλυση μου για το εξή. Θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο παίζεται καλύτερα όταν ο διαιτητής ε, δεν σφυρίζει κάθε πέντε λεπτά για το παραμικρό προκειμένου να υπάρχει ένα όμορφο παιχνίδι. Με την οικονομία μπορεί να υπάρχει μια όμορφη, ρέουσα οικονομία και μπορεί να είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό. Όπως αυτό συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Συμφωνείτε? Η κυρία Φαγιόν, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Εγώ ίδια δεν παίζω ποδόσφαιρο. Όμως στον αθλητισμό υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και γι' αυτό θα ευχόμουν να μπορούσαμε στην Ευρώπη να μπορούσαμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές ε, αθλητισμού και για αυτή την ε, παρομοίωσή σας για το τι μπορούμε να κάνουμε για την οικονομία, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη μπορεί αυτό το παράλληλο ο να ισχύει. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο κύριος Τάνκ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και φυσικά για να μπορούμε να παίξουμε σωστά θα πρέπει να υπάρχουν ισότιμοι όροι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι φιλόδοξη. Αυτό μου αρέσει γιατί χρειάζεται πραγματικά προκειμένου να αδράξουμε αυτήν την τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη. Είναι λοιπόν, ε, υπάρχει αυτό το ερώτημα. Θα δείξει αυτή τη φιλοδοξία για το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρία θέματα έχω να θέσω ε, ως ερώτημα. Καταρχάς, καλύτερη ρύθμιση δεν ε, μπορεί να υποβιβαστεί σε μία συζήτηση για κάθε μικροκανονισμό. Η καλύτερη ρύθμιση σημαίνει μία καλύτερη Ευρώπη πιο κατανοητή σε όλους. Η νομοθεσία για το περιβάλλον χρειάζεται προκειμένου να υπάρχει βιώσιμη οικονομία και αυτό συμφέρει τους πάντες. Και χαίρομαι που άκουσα ότι μπορούμε να περιμένουμε νέες προτάσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και για την κυκλική οικονομία φέτος ακόμα. Κατά δεύτερον, το LuxLeaks κατέδειξε ότι κάτι πάει στραβά με το πρόγραμμα της Ευρώπης. Ζητείτε λοιπόν νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πιο μεγάλο με πιο πολύ ανοιχτό χαρακτήρα, εκθέσεις αναχώρα, ε, μαύρους καταλόγους, μαύρες λίστες και με πιο πολύ ρύθμιση προκειμένου οι μονομερείς αυτοί φορολογικές, οι μονομερείς φορολογικές ε, ρυθμίσεις να καταργηθούν. Και κατά τρίτον, ο κύριος Γιούγκερ μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε τριπλό α. Αυτό δεν γίνεται χωρίς ε, πλήρης αναρρύθμιση, μεταρρύθμιση Τη ε, σχετικής νομοθεσία. και αυτό χρειάζονται. Σα ευχαριστώ. Διακόπτει ο πρόεδρο, Η κυρία Αρένα για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί περί των ουσιοδών. Η κοινωνική προστασία για μένα είναι θεμελιώδη δικαίωμα στην Ευρώπη. Στο πρόγραμμα εργασία εννοείται ότι το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια τη κινητικότητα των εργαζομένων και ότι η λύση θα ήταν η καταπολέμηση των καταχρήσεων. Αλλά κύριοι και κυρίες επίτροποι, το κοινωνικό τόπινγκ κάτι παραπάνω. Είναι μια επίθεση κατά του ευρωπαϊκού κοινωνικού συστήματος. Ε, δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ εργαζομένων και κανεί εργαζόμενο δεν κερδίζει, κανεί δεν προστατεύεται καλύτερα, κάτι ανεργία μειώνεται, ε, προστατεύεται λιγότερο και τον εκμεταλλεύονται. Και δεν κερδίζουν μικρομεσαίε επιχειρήσει. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει προσπαθούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που σήμερα κρεοκοπούν στην Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Γιούνκερ, ούτε εσεί ούτε εγώ ε, δεν εξελέγημεν για να καταστρέψουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων ή να καταστρέψουμε τον ιστό των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι προτεραιότητα η αναθεώρηση οδηγία για τι αποσπάσει, αλλά από όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε η κοινωνική προστασία στην Ευρώπη να είναι μια προτεραιότητα πράγματι. Δεύτερο σημείο που αφορά την μητρική άδεια. Χαίρομαι που βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους αυτή τη θεματική τη βάζει στο, στο θεματολόγιο τη. Θα πρέπει όλοι να απομισθούν τι ευθύνε τη. Και λέω ότι έξι μήνε δεν είναι πολύ. Μία εγκυμοσύνη κανονικά είναι εννέα μήνε. Ελπίζω να μα δώσετε το χρόνο να φτάσουμε τελικά σε μία λύση. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Ούτσιλι, ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ. Με το μικρόφωνο παρακαλώ. Sorry. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ελπίδες ε, και υπεψηφίσαμε την υποψηφιότητά σας πριν από κάποιες εβδομάδες επειδή πιστεύαμε ότι θα προαγάγατε την οικονομία, θα είχαμε ανάπτυξη και το πρόγραμμά σας σα συνεισέφερε να μειωθεί η ανεργία. Ξέρετε ποιος τομέας είναι εκείνος που συνεισφέρει περισσότερο ώστε πραγματικά να διασφαλίζουμε καλές θέσεις εργασίας ε, και να έχουμε επενδύσεις είναι ο τουρισμός και ο τουρισμός ακριβώς ε, με ούτε λέξη δεν παρουσιάζεται στο πρόγραμμα εργασίας σας. Όταν όμως ε, κάνουμε λόγο για μια ανταγωνιστική ολοκληρωμένη Ευρώπη πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό τον τουρισμό. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία πρέπει να στραφούμε στον τουρισμό. Πρέπει να δούμε ότι τα έσοδα, 50% όλα των εσόδων στην Ευρώπη προέρχονται από τον τουρισμό συνολικά. Θα ήθελα λοιπόν να, να σας προσφέρω να σας βοηθήσουμε. Ήμουν προηγούμενας κάτω παρελθόν ε, ε, υφυπουργός όσον αφορά θέματα τουρισμού και πάμπολη σε σχέση με τους ευρωβουλευτές σας στη διακομματική ομάδα για τον τουρισμό παρενέβησαν και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε και αυτός ο τομέας να αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας σας ο τουρισμός από την Ουγγαρία την προηγούμενη εβδομάδα σας απέστειλα μια επιστολή κύριε Πρόεδρε Ιούνκερ και ανέφερα σε αυτήν ότι μέσα στο πλαίσιο μέσα στο ε, προεκλογικό πρόγραμμα ε, ε, υπήρξαν παραβιάσεις ε, αρχών και νομοθεσίας. Δεν μου δώσατε όμως απάντηση σε αυτή την επιστολή μου. Μόνο μια δήλωση απεστάλλει προς τον Ουγγρικό τύπο που διαβιβάστηκε σε αυτόν. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη θετική μας συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ούτσελη. Και στη συνέχεια με τον κατάλογο των αγοριτών που ολοκληρώσαμε ακολουθεί η διαδικασία Catch the μια και ολοκληρώθηκε η προηγούμενη έχουμε πάνω από 20 αιτήματα να παρέμβουν ευρωβουλευτές έχουμε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο λοιπόν και τη διακριτική ευχέρεια ε, την ε, άσκησα ώστε να μπορέσω να ε, κατανείμω τον χρόνο με τον δικαιότερο τρόπο σε σχέση με τα αιτήματά σας. Θα σας πω τα ονόματα εκείνων που θα παρέμβουν. Speeches, one minute. And there will be eight of these. οκτώ από θα Mr. Siekierski, Mr. Tarabella, Mr. Seraf Santos, Mr. Marias Notis, Mr. Faria, Mr. Senra Rodriguez and Mr. Castaldo Uh, Μπορεί να υπάρξει διαφορετική σειρά, αλλά από αυτούς θα υπάρξουν οι παρεμβάσεις. Ο κύριος Λαβία πρώτος, παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο παρέμβαση. Can I start? Ξεκινήσω. Madam Senator Rodriguez. Κύριε Rodriguez. Right. Please. Να μπείτε στον κατάλογο, εντάξει, ορίστε. Κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ, Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, σαν Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου και εν ονόματι των συντονιστών όλων των πολιτικών ομάδων, δηλώνω την πλήρη ανικανοποίησή μου, την προσωπική και των συναδέλφων, για την απόσυση του νομοθετικού πακέτου για την κυκλική οικονομία και για την ανάλογη πρωτοβουλία για το Air Quality Package. Ακούσαμε τη νέα σας πρόταση αυτό που μόλις βγήκε από τον τύπο για τις, προ... για τις προτάσεις τις βελτιωτικές που θα κάνετε. Περιμένω να τις δούμε. Αν μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εξηγήσει σε τι θα είναι βελτιωτικέ οι νέε προτάσει, θα το εκτιμούσαμε να τα ακούσουμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σα καλέσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντο επανειλημμένα και περιμένουμε ακόμα την επίσκεψή σα. Είναι σαφέ ότι δικαιολογήθηκε η απόσυση του πακέτου απλώς βάσει του εξής. Δηλαδή, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει συμφωνία διαθεσμική. Και πριν έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε το μέτρο, θεωρήσαμε ότι ήταν γελίο αυτό, τουλάχιστον. Σε Σας ευχαριστώ. κ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει μετά από δύο ώρες συζητήσεων να φτάσουμε να μιλήσουμε για τη γεωργία 38% του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Καλύτερο νομοθετή είναι ήδη ξεκίνησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα χαρτοφυλάκιο που είναι η διανομή των απορροκυπηστικών, των οπών και των, ε, για, της βοήθειας τα σχολεία. Απλουστεύοντας την όλη κατάσταση να είναι πιο προσβάσιμα τα προϊόντα και να υπάρχει και εκπαίδευση γύρω από τα τρόφιμα που είναι θεμελιώδες. Είμαι συγκητής του Κοινοβουλίου, η έκθεσή μου κατετέθη ήδη, είναι στη μετάφραση και θα ήταν κρίμα που δεν την ψηφίσαμε. Η προσοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να παραμείνει αυτό. Θα ήθελα διευκρινήσει και ο κανονισμό για την βιολογική γεωργία. Η παραγωγή τη βιολογική γεωργία θέλουν προστασία, υπάρχουν ψευδή προϊόντα, έχουμε εισαγωγή 30% όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα στον, στην Ευρώπη. Ζητούν η παραγωγή προστασία. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αποσύρει το σχέδιο κανονισμό. Τι να πούμε για του πόρου, υπάρχουν προσδοκίε, είναι κάτι που αναβάλαμε σαν θέμα. Ποια είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του πόρου. Θα ήταν θεμελιώδε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σήμα στο γενικό τομέα που έχει μεγάλη ανάγκη που κάτι τέτοιο σήμερα. Κύριε Γιούνκερ, εκπλήσωμαι που σας ότι είχατε πάει στην Αθήνα για να στηρίξετε επιτόπου τους μνημονιακούς πολιτικούς σας φίλους. Μια και ο κύριος Μοσκοβισή που στείλατε στην Ελλάδα τα έχει κάνει θάλασσα. Κύριε Γιούνκερ, με τις πρόσφατες δηλώσεις σας εκφράσατε πολιτική προτίμηση σε συγκεκριμένους γνώριμους σε εσάς, όπως είπατε, πολιτικούς εν ώψη των επικείμενων γενικών εκλογών στην ελλάδα. ποιο νομίζετε ότι είστε κύριε Γιούνκερ, ο νέο ανθίπατο των αθηνών; ποιο σα έδωσε το δικαίωμα να παρεμβαίνετε ομά στην εσωτερική πολιτική κατάσταση τη ελλάδα; τελικά είστε πρόεδρο τη επιτροπή ή εκπρόσωπο τη τρόικα και των δανειστών. συμμαζευτείτε λοιπόν κύριε Γιούνκερ, τηρήστε την πολιτική ουδετερότητα που σα επιβάλλει η συνθήκη. πάρτε το απόφαση κύριε juncker θα το πιείτε το πικρό ποτήριο και εσείς και η μνημονιακή πολιτική σας φίλη στην ελλάδα γιατί ο ελληνικός λαός θα σας στείλει μήνυμα στις επόμενες γενικές εκλογές. ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Αντιπρόεδρε. Κάνουμε λόγο για το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 εσείς όμως ε, την ομοθεσία για το περιβάλλον της διαγράφετε, της ακυρώνεται για την ανακυκλούμενη οικονομία επιπλέον θα υπάρξει στραγγαλισμός αυτό, λόγω αυτής της πολιτικής θα μειωθεί, ε, αντί να μειωθεί η ρήπανση του αέρα, αντί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής ε, και ε, να λάβουμε υπόψη την ανακύκλωση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα γίνει τίποτα από αυτά. Και ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Τίμερμανς, όλα αυτά τα κυρώνει. Κύριε Γιούνκερ, γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφορα κράτη-μέλη και η Γερμανία και η Γαλλία που ζήτησαν την Επιτροπή να διατηρηθούν αυτές οι δύο οδηγίες. Τι θα γίνει. Υπάρχει εδώ λοιπόν μία αντιπαράθεση σε σχέση με τον κύριο Τίμερμανς και τον Επίτροπο για το Περιβάλλον που είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα επέτρεπε να καταργηθούν αυτές οι δύο περιβαλλοντικές οδηγίες. Ευχαριστώ. Σενιόρα Σένρα Ροντρίγκες. Σε ευχαριστούμε. Ροντρίγκες παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γιούγκερ. Μία από κάθε τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται ανδρική βία. Δεν είδα τίποτα από τους προτεραιότητες εργασίας σας για το 2015 να καταπολεμηθεί αυτή η μάστιγα. Η γεωργία, η αλληλεία, οι δυο δηλαδή αυτές βάσεις ε, της ε, ε, επισητιστικής κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι για αυτά δεν είδα τίποτα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μηδέν, τίποτα για αυτές. Φτώχεια, πείνα, κοινωνικός αποκλεισμός. Ούτε για αυτά είδα τίποτα στι προτεραιότητε για να καταπολεμηθούν αυτά τα θέματα. Πρόσβαση στη στέγαση ή να αποφύγουμε να χάνουν τη στέγη του στο διαμέρισμά του χιλιάδε πολιτών κάθε μέρα. Πάλι μηδέν στι προτεραιότητε σα. Τίποτα όσον αφορά την επισφαλή εργασία. Τίποτα όσον αφορά την απώλεια εργατικών δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων που κάθε μέρα αυξάνεται η απώλεια αυτή. Τίποτα για τι βασικέ υπηρεσίε όπω ε, το δικαίωμα για την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες. Ε, τι είναι όλα αυτά λοιπόν, πώς μπορούν να δικαιολογηθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια... Καστάλτο, παρακαλώ. Εδώ και χρόνια ο Παύλο Μπορσελίνο, ο μεγάλο άντρα, έλεγε ότι η πολιτική και η μαφία είναι δύο εξουσίε που ζουν από τον έλεγχο τη ίδια επικράτεια. Ή κάνουν πόλεμο ή τελικά κάνουν συμφωνία πολύ συχνά νικάει η συμφωνία. Το ξέρουν πολύ καλά οι τίμοι, οι πολίτε τη πόλη τη Ρώμη, που συγκλονίστηκαν από μια έρευνα που δείχνει πιο σοβαρά πορίσματα. 37 συλλήψει, πάνω από 80 διοκόμενοι, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, συνεταιρισμοί, δημοσιογράφοι, στατιωτικοί, επιχειρηματίε. Αυτή είναι η μαφία. Αυτή είναι, αυτό είναι το οργανωμένο έγκλημα που είναι και όλο πιο παράτολμη. Όταν παρουσιάσετε το πρόγραμμά σα, Πρόεδρε, λέτε ότι η καταπολέμησή του είναι μια ευρωπαϊκή ευθύνη. Είναι η ώρα να περάσετε από τα λόγια στι πράξει. Η πρόταση κατά τη ανακύκλωση είναι κάτι χρήσιμο, αλλά δεν αρκεί. Αν δεν έχουμε ε, αν δεν γίνεται ε, συνεταιρισμό σε μαφιόζικες ομάδε, αν δεν καταδικάζεται επαρκώ, αν δεν σταματήσουν οι φορολογικοί παράδεισοι, ε, αν δεν υπάρξουν ε, τιμωρίε στον αφορά τις παραβιάσεις κάτω του περιβάλλοντος, τελικά θα επικρατήσει σιωπή. Ο μαφιόζο δεν μπορεί να είναι ένα άτομο που λέμε ότι δεν υπάρχει ε, και άτομα άλλα δεν το γνωρίζουν. Η σιωπή των ευρωπαϊκών θεσμών σκοτώνει. Η σιωπή είναι μαφία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σικέρσκι. Έχετε το λόγο. Πρέπει να σε ευχαριστήσουμε, Πρόεδρε. Ο κύριος Τίμερμανς είπε ότι αν κάτι δεν αναφέρθηκε, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το κάτι δεν είναι σημαντικό. Ε, από αυτό συνάγω ότι οι προτεραιότητες για το 2015 θα είναι πιο πολύ αριθμές. Όμως, παραμένει γεγονός ότι ασχολούμεθα με ένα θέμα, το ότι ασχολούμαστε με ένα θέμα δεν σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας θα στεφτούν από επιτυχία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραδείγματο χάρη οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις, οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, το ρωσικό εμπάργκο, οι ασθένειες ε, όσον αφορά οι των χείρων. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι η βιολογική παραγωγή και τα σχολικά προγράμματα είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα αλλά και σημαντικότατα από πλευράς κοινωνικής. Για να συνοψίσω, πιστεύω ότι αυτά τα προβλήματα δεν θα πρέπει να εγκαταληφθούν, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις προτεραιότητές σας για το 2015. Ε, συμφωνώ μαζί σας και διακόπτει ο Πρόεδρος. Σάντος, παρακαλώ. Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προληπτικά να δράσει για τον γαλακτοκομικό τομέα σε σχέση με το, τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις που θα τερματιστούν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες αυτός ο τομέας. Πολλές φορές σε ζώνες όπου δεν υπάρχει άλλη οικονομική δραστηριότητα. Προέρχομαι από τις Αζόρες που συμμετέχει και συνεισφέρει σε τεράστιο ποσοστό για τον γαλακτοκομικό τομέα και υπάρχει πραγματική ε, θα έλεγα κάλυψη των αναγκών μας με τη καλύτερη τεχνολογία και μια καλή ε, διαχείριση της προσφοράς ε, όσον αφορά την απόσβεση επέ επενδύσεων Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει την πολιτική βούληση ώστε να μπορούν να βρεθούν λύσεις βιώσιμες για την ρύθμιση αυτής της αγοράς γαλακτοκομικών για να μπορέσουν οι διαφορετικές αλλαγές να επιτευθούν και να μπορέσει πραγματικά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και σε σχέση με την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι η κατεξουσία πράξης όσον αφορά τον τομέα της θάλασσας θα μπορέσει να αναφερθεί για τους τομείς που αναφέρονται και όχι για κάποιους τομείς βραχυπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Uh, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος τώρα κύριος Τίμερμανς ε, θα λάβει τον λόγο που είναι αρμόδιος για το καλύτερο νομοθετικό ε, έργο θα λάβει τον λόγο για πέντε λεπτά. Έχετε λοιπόν πραγματικά την ευκαιρία να κάνετε αυτά τα οποία διακηρύτετε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και είναι καινούριο για μένα να με τις απόψεις σας και σε σχέση με την οικονομία κρατών μελών και την κρίση που, ε, στην οποία καταλήγει κανείς ε, για την... Έχω μικρή πείρα, λίγη πείρα σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο, μαθαίνω όμω ταχύτατα. Ήμουν βουλευτή στο Εθνικό Κοινοβούλιο επί πολλά χρόνια. Έξι φορέ έχω επανεκλεγεί και γνωρίζω πώ εργάζεται κανεί σε ένα Εθνικό Κοινοβούλιο. Τώρα πρέπει να συνηθίσω πώ μπορεί κανεί να εργάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο που είναι διαφορετική περίπτωση. Για παράδειγμα, θα ήθελα να είχα απαντήσει στον κύριο Φάρατζ, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα να αναμένει την απάντηση, να μπορεί να περιμένει να δοθεί απάντηση. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν έχω συνηθίσει ακριβώ το γίνεται γίνονται τα πράγματα, αλλά έτσι γίνονται εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεύτερον, ένα έγγραφο διέρευσε την προηγούμενη εβδομάδα και ε, ο πρόεδρος και εγώ ανησυχήσαμε γι' αυτό διότι αυτό δεν μας βοηθά να εργαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργείται δίνεται μεγάλη διάσταση από τον τύπο σε αυτά και εσείς αντιδράτε και όλας και πολλοί από εσά αναφέρθηκαν σε αυτό το έγγραφο που διέρευσε αποφάσισα με την κοινοβουλευτική μου πείρα να μην αντιδράσω θα μπορούσα αμέσω να είχα πει δεν είναι αυτό, δεν αληθεύει δεν είναι αυτό το οποίο κάνουμε είναι τελείως διαφορετικό εμείς άλλες αποφάσεις λαμβάνουμε για το τι θα κάνουμε. Αλλά ε, λόγω σεβασμού στο Κοινοβούλιο δεν αντέδρασα. Ήθελα να παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασία ε, τη Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και όχι στον τύπο. Τουλάχιστον λοιπόν με ένα χέρι δεμένο πίσω από, το χέρι, από τη, τη, την πλάτη του αμήνεται κανεί ε, όταν υπάρχουν τέτοιε διαρροέ ε, και όταν γίνονται τέτοιε τοποθετήσει για τέτοιου είδου έγγραφα. Με ρωτάτε αν δείχνω τον σεβασμό που απαιτείται στο Ευρωκοινοβούλιο παρουσιάζοντα το πρόγραμμά μα εδώ. Και να το λάβετε υπόψη λοιπόν και παρακαλώ να ακούτε αυτά τα οποία λέω και να αντιδράτε σε αυτά τα οποία λέγω εγώ και όχι σε αυτά τα οποία αναφέρεται μια, ε, ε, ένας ψήθυρος ή μια φήμη στην οποία αναφέρονται δημοσιογράφοι την οποία εσείς ε, διαβάσατε ως είδηση και σε αυτήν αντιδράτε. Ε, λοιπόν, πραγματικά αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι και όπως το είπα σαφώς για το περιβάλλον θα κάνουμε, θα διατηρήσουμε ε, προγράμματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και υφίστανται. Θα επανεξεταστεί το πρόγραμμα για τα απόβλητα, αλλά θα ολοκληρωθεί σε σχέση με την ανακυκλούμενη οικονομία και θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν κέρδη από τις ευκαιρίες που θα προσφέρει το πρόγραμμα Juncker για επενδύσεις σε αυτή την ανακυκλούμενη οικονομία. Δεν θα μειώσουμε τον πύχη όσον αφορά τις φιλοδοξίες μας. Δεν θα τις υποβαθμίσουμε όσον αφορά την διασφάλιση καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα για τους Ευρωπαίους. Δεν θα υποβαθμίσουμε, επαναλαμβάνω, της τις προσδοκίες και τι απαιτήσει. Θα υποβάλουμε όμως προτάσεις και θα τις καταθέσουμε στο τραπέζι και ό,τι υπάρχει και είναι περιττό και θεωρούμε ότι μπορούμε να πράξουμε καλύτερα θα το επανεξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της ε, ως ε, ανεξάρτητο όργανο υποβολής προτάσεων με δική της πρωτοβουλία για να ληφθεί απόφαση για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτό είναι ο ρόλος μας και αυτό θα κάνουμε. Αλλά με μια θετική μερίσια διάταξη ω θεματολόγιο και όχι υποβαθμίζοντας ε, τις προδιαγραφές μας. Και για τα κοινωνικά θέματα είναι τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγουμε αυτά τα πράγματα στον κοινωνικό τομέα και να σημειωθεί πρόοδο όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την κινητικότητα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την κινητικότητα, να καταπολεμήσουμε όμω τι καταχρήσει, διότι οι καταχρήσει υπονομεύουν την ελευθερία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση για του εργαζόμενου να χρησιμοποιήσουν ευκαιρίε σε άλλα κράτη-μέλη να βρουν εργασία εκεί και να απασχοληθούν εκεί, αν αυτό είναι διαθέσιμο σε ευκαιρία. Πώ θα τα κάνουμε όλα αυτά. Θα έχουμε μια ευρύτερη βάση για να ενημερώνουμε για να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι θα επικαιροποιήσουμε τους κοινωνικούς κανόνες και κανονισμούς για την απόσπαση εργαζομένων ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιείται ώστε να υπονομεύονται ρυθμίσεις και διατάξεις και όπως το προαναγγείλαμε θα υπάρξει μια στοχοθετημένη αναθεώρηση για την οδηγία απόσπασης εργαζομένων θα ξεκινήσει το 2015 ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο και το έχουμε αναγνωρίσει. Μιλήστε με αυτούς που εργάζονται στις αναφορές και θα δείτε. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες μας. Και όταν κάνουμε λόγο λοιπόν για θέσεις των γυναικών και αυτό έχει τεράστια σπουδαιότητα. Δεν κάνουμε λόγο απλά και μόνο για το τι είναι ηθικά σωστό και δίκαιο. Εγώ ως πατέρας οπωσδήποτε δεν μπορώ να δεθώ οι δυο μου κόρες να βρεθούν σε χειρότερη θέση στην αγορά εργασία ή στην κοινωνία από ότι οι δυο μου γη. Κάτι τέτοιο θα ήταν απόλυτα παράδεκτο για μένα. Όμω υπάρχουν και σαφέστατοι οικονομικοί λόγοι για του οποίου δρούμε. Διότι υπονομεύεται η οικονομία τη Ευρώπη και τα συμφέροντά τη όταν δεν υπάρχει ένα ισοδίκαιο, ισότιμο πλαίσιο δραστηριοποίηση για όλου. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ για όλα αυτά. Και για την πρόταση για οδηγία όσον αφορά την μητρική άδεια, ε, για πολλά κράτη-μέλη ήδη είχε ήδη παρακαμφθεί από την πραγματικότητα σε αυτά τα κράτη-μέλη. Επί 8 χρόνια βρισκόταν επί τραπέζης, είχε τροχοπεδηθεί, είχε προχωρήσει η κατάσταση παραπέρα. Θέλουμε εμείς να βελτιώσουμε όμως συνολικά την κατάσταση και μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν με αυτή την πρόταση. Δείξτε μας άλλα θεσμικά όργανα που μπορεί να γίνει και θα το κάνουμε. Όμως τα πράγματα αν δεν προχωρήσουμε δεν βελτιώνουν την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και αν δεν βελτιώνεται η κατάσταση θα λάβουμε άλλα μέτρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, για να βελτιωθεί, να σημειωθεί βελτίωση και πρόοδος. Φυσικά ο κύριος Φάρατς αν υπήρχε, ήταν ακόμα εδώ, θα του έλεγα ότι σε ένα σημείο συμφωνώ μαζί του. Και είναι καλό να συζητούμε πράγματα επί των οποίων συμφωνούμε. Θα του έλεγα ότι έχει δίκιο όταν αναφέρει ότι υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση γραφειοκρατική πανευρωπαϊκά εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρέπει επιτέλου να κάνουμε κάτι, να ανακουφίσουμε αυτή την επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν υπάρχει περάσει αυτή η επιβάρηση αν ανακουφιστούν ταχύτατα θα προσλάβουν ένα-δύο επιπλέον εργαζόμενους και αυτή θα είναι μια άμεση συνεισφορά για να καταπολεμηθεί η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μια φορά επιτέλους πίστευα ότι ο κύριος Φάραζε είχε ένα φιλευρωπαϊκό πνεύμα. Νομίζω ότι είναι γενικότερη η εντύπωση, αυτό το μάθαμε από το UKIP ότι καμιά φορά λέει κάτι που είναι σωστό. Θα ήθελα όμως να εμπλακεί αυτή τη συζήτηση και ο ίδιος Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη τελικά όλοι μια τελική παρατήρηση, διότι αναφέρθηκε από αρκετούς, από πολλούς. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα και επειδή ένα, όταν ένα θέμα είναι σημαντικό δεν σημαίνει ότι αμέσως η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει άμεσα. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην αγορά εργασίας, αν θέλουμε να βελτιώσουμε τα κοινωνικά θέματα στα κράτη-μέλη, αυτό δεν θα γίνει μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ρόλο να διαδραματίσει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι εξίσου σημαντικό τα κράτη-μέλη να αναλάβουν μέτρα και πρωτοβουλίε για να προχωρήσουν όλα αυτά. Γι' αυτό θα πρότεινα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, και το Κοινοβούλιο να καταβάλουν προσπάθεια να πείσουν το Συμβούλιο για όλα αυτά. Πολλά από αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο θα πρέπει να εμπλακούν, να δράσουν για να μπορέσουμε να προαγάγουμε αυτά τα θέματα. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προετοίμασε το πρόγραμμα εργασίας σας το παρουσίασε σήμερα και όσον αφορά εμένα προσωπικά είναι η έναρξη ενός διαλόγου μαζί σας. Δεν είναι η τελεσίδικη τελική καθοριστική λέξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα φουγκραστούμε τις απόψεις σας προσεκτικά ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης και αυτό το οποίο θέλει η Επιτροπή Juncker όταν εξελέγει και δήλωσε ότι επιθυμεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα για να κλείσετε τη συζήτηση ο Πρόεδρος Γιούγκερ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δρούμε. Παρέσει συνεδρίαση των Προέδρων των Επιτροπών όπου όλα υπόθηκαν και όπου δεν υπήρχε σύγχυσης. Ο Φαν Τίμερμαν και εγώ παρέστημε λοιπόν στη διάσκεψη των Προέδρων σήμερα και έχω την εντύπωση ότι αυτή η συνεδρίαση ε, δεν λήφθη υπόψη. Θέλαμε να παρουσιάσουμε σε εσά το πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήθελα να την παρουσιάσω και στον τύπο. Δεν σχολιάζουμε αυτά που υπόθηκαν. Ε, Uh, Δεν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά στο Κοινοβούλιο. Παρακαλώ να το αφαιρέσετε αυτό. Okay. Συνεχίστε, Πρόεδρε Γιούνκερ. Κατανοώ λοιπόν τις διάφορες ομιλίες που γίνονται σε κανονική γλώσσα. Δεν χρειάζεται να μου δείχνετε σύμβολα και σημαίες. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τα πράγματα και καταλαβαίνω. Θα ήθελα να σας να πω ενώπιος σας ότι θα ήθελα με τον Πρόεδρο και διάσκεψη των έχω μια συνεδρίαση για τη μέθοδο εργασία όσον αφορά την παρουσίαση και συζήτηση των προγραμμάτων εργασία. Είναι απογοητευτικό σήμερα αυτό και για σας και για μας. Δεν θέλουμε να... Θα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορές λοιπόν και κανόνες για να μην έχουμε συνέχεια διαχείριση της απογοήτευσης. Να επανέλθω σε κάποια σημεία για να τα διευκρινίσω. Ακούμε το Κοινοβούλιο, ακούμε το Συμβούλιο. Και βλέπω ότι κανείς δεν υπογράμμισε το βασικό κανένα της διοργανικής ευγενίας. Και ο Τίμερμανς και εγώ αποσύραμε από τον κατάλογο των πρωτοβουλειών που εκκρεμούν όλα τα προγράμματα που βρήκαν αντίσταση καμιά φορά πολύ μεγάλη από το Κοινοβούλιο και αντίδραση του Κοινοβουλίου. Πάκτα ε, out. Budendienst και άλλα στοιχεία ε, που βρήκανε πολύ ε, ισχυρή αντίσταση του Κοινοβουλίου απεσήθησαν το πρόγραμμα εργασίας. Κάνατε λάθος που δεν το αναφέρατε. Αν παρουσιαστήκαμε μπροστά σας λέγοντας ότι όλα είναι επιτάπητος και οι προτάσεις εκείνες που είχατε απορρίψει, αν σας λέγαμε αυτό, θα κάναμε αυτό που έκαναν άλλοι. 130 νέες προτάσεις. Όλα παραμένουν επιτάπητος, δεν αποσύρουμε τίποτα. Θα έχουμε 130 νέες προτάσεις. Θα χειροκροτούσατε. Κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου και θα το κάνουμε και του χρόνου. Παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα για το 2015, τον επόμενο χρόνο. Παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα για το 2016. Όσον αφορά τη φορολόγηση όλα υπόθηκαν και όλα θα γίνουν. Αυτό αναφέρθηκε στην προεκλογική εκστρατεία και στην παρουσίαση των προσανατολισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκαν. Θα γίνουν αυτά. Μιλήσαμε πολύ για διαφάνεια. Ε, καμιά φορά πιάνει μανία αυτή την αίθουσα με τη χρήση αυτής της λέξης. Και εγώ και ο Φραν Τίμερ μα τελευταίε εβδομάδε εργαστήκαμε. Κάναμε πρόταση για τη διαφάνεια εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επίτροποι, τα γραφεία, γενικοί διευθυντέ θα πρέπει να ενημερώσουν το κοινό όσον αφορά τη φύση και ταυτότητα ε, αυτών των διαφόρων συναντήσεων και εκείνων που είδανε. Δεν είπα ότι το κοινό που είπα κάνει το ίδιο. Κάντε το αν θέλετε. Κάντε το. Ας είστε εξίσου ε, ε, καλεί όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψηφίστε ένα ψήφισμα και να πείτε ότι θα κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την Ελλάδα, εγώ δεν καταλαβαίνω ελληνικά. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγραψαν οι ελληνικές εφημερίδες. Όταν αναφέρθηκα στους εξτρεμιστές στην Ελλάδα, δεν υπερασπιζόμουν την άκρα δεξιά. Ε, η ιδέα δεν μου πέρασε το μυαλό ότι θα μπορούσατε να είστε εξτρεμιστές. Δεν κατανοώ λοιπόν γιατί η αριστερά η ελληνική υπερασπίζεται την άκρα δεξιά. Εγώ μισώ την άκρα δεξιά, μισώ την άκρα δεξιά, την απεχθάνομαι. Και πρέπει να το πω. Και έχω το δικαίωμα κατά τα λοιπά, είμαι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ερχόμενο στο Στρασβούργο, ότι ξαφνικά ε, έχασα τις πεπιθήσεις μου. Μπορώ να πω τα πράγματά μου. Το λέω συχνά στη Γαλλία και στο Βέλγιο, λέω πράγματα που δεν ε, ευχαριστούν ούτε την εξουσία ούτε την αντιπολίτευση. Ε, λοιπόν, η Ευρώπη είναι πολιτική Ευρώπη και επίση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολιτική. I will convey your concerns about... Uh, Να εκφράσω μια ανησυχία για τη διαδικασία και για την ε, διαφάνεια ε, στην διάσκεψη των Προέδρων. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην επόμενη σύνοδο του Ιανουαρίου. Ε, Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Γιούγκερ και τώρα συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τον προπολογισμό. Πρωτού όμως περάσουμε στη συζήτηση για τον προπολογισμό να αναφέρω ότι σε σχέση με τη σύσταση της απόφασης από την Επιτροπή Ίντα να μην εκφραστούν ενστάσεις για την ε, πράξη καταξιοδότηση που αναφέρθηκε χθε στην χθεσινή συνεδρίαση δεν εκφράστηκαν σχετικέ ενστάσει εντό 24 ώρων και σύμφωνα με τον κανόνα 105 παράγραφο 4 εγκρίνεται η σύσταση αυτή. Θα δημοσιευτεί με τα εγκεκριμένα κείμενα αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου του 2014. Να ενημερώσω επίση το Κοινοβούλιο ότι σύμφωνα με τον κανόνα 231 παράγραφος 4 δεν εκφράστηκε έτοιμα να ψηφιστεί το